Morning, ladies and gentlemen. I like, I want to start, but normally we start with the rapporteur. Λοιπόν, ας αρχίσουμε σήμερα. What shall I do? Is there possible... Θα πρέπει να ξεκινήσουμε με τον εισηγητή, αλλά δεν τον έχω δει ακόμη, οπότε ίσως να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σήμερα έχουμε πάλι πολύ φορτωμένη ημερήσια διάταξη, πολλά θέματα που πρέπει να συζητηθούν σημαντικά και μέχρι τις 10 η ώρα που θα αρχίσουν οι ψηφοφορίες έχουμε να κάνουμε δύο πράγματα. Θα ήθελα να αρχίσω με το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης και να δώσω στην συνάδελφο εισηγήτρια το λόγο στη Ρωμάνα Ιόρνταν Σίσλικ. Παρακαλώ. Herbert, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως όλοι γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2010 μας υπέβαλε μία πρόταση για οδηγία του Συμβουλίου για τη διαχείριση των ραδιονοργών αποβλήτων και αναλωμένων καυσίμων. Η οδηγία αυτή αποτελεί την εξακολούθηση του έργου της Επιτροπής με την οδηγία του 2003, όπου η Επιτροπή είχε υποβάλει κοινή πρόταση για δύο οδηγίες, την οδηγία ε, πυρηνική ραδιονεργή ασφάλεια και την οδηγία για τη διαχείριση των αποβλήτων. Εκείνο το, πακέτο, εκείνο το τη δέσμη μέτρων την είχαμε ονομάσει πυρηνικό, το ραδιενεργό πακέτο. Το πακέτο περί ραδιενεργών αποβλήτων. Την οδηγία αυτή την είχαμε Εξετάστηκε και προηγουμένω στο Κοινοβούλιο και στο τέλο τη προηγούμενη θητεία είχαμε εγκρίνει και την τρίτη οδηγία. Τώρα έχουμε επιτάπητο πρόταση οδηγία για τη διαχείριση των αλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων. Γιατί όμω απορρίφθηκε η οδηγία το 2003. Η βασική επίκριση ήταν ότι δεν έλαμβανε υπόψη την αρχή τη επικουρικότητα. Υπήρχαν και άλλε αποκλήσει απόψεων, διότι Κάποιοι έλεγαν ότι οδηγία ορίζει ένα κοινό σύστημα επενδύσεων, Όμω τα κράτη-μέλη θεωρούσαν ότι οι προποθέσει για τη χρηματοδότηση τέτοιων δραστηριοτήτων παρά ήταν αυστηρέ. Και κάτι ακόμη. Δεν είχε τύχει θετική αποδοχή στο γεγονό ότι οι οδηγίε όριζαν πολύ αυστηρέ προθεσμίε για την ε, δημιουργία των εγκαταστάσεων διαχείρισης. Η ημερομηνία λήξη, το όριο ήταν το 2018. Ήταν πολλά τα κράτη-μέλη που δεν θα προλάβαιναν να τηρήσουν αυτή την προθεσμία. Επίσης και για τις επιθεωρήσεις υπήρχε πρόβλημα. Επιθεωρήσεις που επέβαλε η Επιτροπή στους εθνικούς ρυθμιστέ, τους ρυθμιστές και ελεγκτές των κρατών μελών. Θα έπρεπε να αναλάβει Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων μαζί με τα κράτη-μέλη, όμω θεωρούσαν ότι εκεί υπήρχε παραβίαση τη αρχή τη επικουρικότητα. Οι προετοιμασίε για την ε, έγκριση λοιπόν του πακέτου δεν πήγαν καλά. Πιστεύω όμω τώρα ότι το συνολικό τοπίο έχει βελτιωθεί. Έχουν γίνει πολλέ συζητήσει μέχρι τώρα και επιβεβαιώνουν ότι η οδηγία για την διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένων καυσίμων είναι αναγκαία. Αυτό ε, το επιβεβαίωσε η Ειδική Επιτροπή, ομάδες εργασίας, ομάδες δράσης που είχαν αναλάβει τη συζήτηση για αυτή την οδηγία. Επιτρέψτε μου τώρα να πω ε, λίγα λόγια για τη μεθοδολογία μας. Θα γνωρίζετε ότι η πρόταση οδηγίας αυτή βασίζεται στη συνθήκη Euratom. Ευρατόμ. Για το λόγο αυτό, περιλαμβανόταν στη διαδικασία διαβουλεύσεων. Το κοινοβούλιο εδώ έχει ρόλο συμβουλευτικό. Εγώ λοιπόν θα έλεγα να ετοιμάσουμε την έκθεσή μας με τις τροπολογίες αν επρόκειτο για έκθεση επινομοθετικής πρότασης. Θα έλεγα η έκθεση να συζητηθεί στις 31 Μαρτίου. Χθε υπέβαλα στους συναδέλφους μου, τους και το χρονοδιάγραμμα όπως το έχω προβλέψει. Προβλέπεται τον Ιούνιο στη δεύτερη Ολομέλεια να γίνει η ψηφοφορία και η Ουγγρική Προεδρία μου ζήτησε παρόλα αυτά να, προλα... να, κάνω λίγο πιο γρήγορα, να κάνουμε λίγο πιο γρήγορα για να γίνει πιο νωρίς η όλη έγκριση. Θέλει η Ουγγρική Προεδρία επί, της δικού τη εξαμήνου να συζητηθεί η πρόταση αυτή και να ολοκληρωθεί και η διαδικασία. Το συζήτησα λοιπόν με του κοιόδη εισηγητέ και με τον πρόεδρο Ρόιλ, τον κύριο Ρόιλ, και θα δούμε κατά πόσον είναι εφικτό η ψηφοφορία στην Επιτροπή Ήτρε αντί για 26 Μαΐου να γίνει στις 9 Μαΐου. Οπότε τότε θα μπορούμε να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια του Ιουνίου σίγουρα. Αυτό βεβαίω σημαίνει ότι θα πρέπει να προβλέψουμε επιπλέον συνεδρίαση τη Επιτροπή ΙΤΡΕ εντωμεταξύ. Προκειμένου να, να προλάβουμε. Ίσως όμως πριν αποφασίσουμε οριστικά να περιμένουμε λίγο ώστε να δούμε πώς θα τοποθετηθούν τα μέλη της Επιτροπής και να δούμε και πόσος χρόνος απαιτείται για να βρεθούν λύσεις εφόσον τα προβλήματα είναι πολύπλοκα. Θεωρούμε ότι ο χρόνος που θα χρειαστεί για τις διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο πρέπει να μας επιτρέψει να έχουμε ε, θετικά αποτελέσματα, να συνεργαστούμε αποτελεσματικά ώστε να κάνουμε και πιο γρήγορα. Ήδη έχει οργανωθεί μια ακρόαση το Δεκέμβριο, οπότε η διαδικασία έχει ξεκινήσει. Τώρα μερικά λόγια για την ίδια την πρόταση οδηγία. Οι στόχοι τη οδηγία αυτή ήταν τρει. Ο πρώτο είναι όλα τα κράτη-μέλη να λάβουν νομοθετικά μέτρα για την διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων. Δεύτερο στόχο, το κόστο. Το κόστο τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων, το οποίο θα πρέπει να αναλάβουν αυτοί που έχουν παράγει τα απόβλητα. Και έπειτα, ε, ένα άλλο θέμα είναι οι δυνατότητε παρέμβαση τη νομοθεσία όπω έχει υλοποιηθεί από τα κρατη Δεύτερος στόχος, ε, τα όσα αφορούν τον θεμετό ανταγωνισμό στην κοινή αγορά ε, ενέργειας. Προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι ο Ριπένον, εκείνος δηλαδή που έχει παραγάγει τα ραδινεργά απόβλητα, κατά την χρήση των πηγών προβλέπει τέτοια μέτρα οικονομικά, τέτοια μέσα οικονομικά που μπορούν μετά να εξασφαλίσουν την ασφαλή διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων. Θα πρέπει έτσι να καλύπτεται από την τιμή του τελικού προϊόντος το κόστος της διαχείρισης, δηλαδή η τιμή της ενέργειας, η οποία πωλείται στην ε, ελεύθερη αγορά. Η τιμή λοιπόν αυτή πρέπει να καλύπτεται από τον υπεύθυνο, η τιμή της απομάκρυσης και από τους διαφορετικούς παραγωγούς ε, και πολιτές ε, προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά. Επίσης μας ενδιαφέρουν τα μέτρα που προβλέπουν υποχρέωση ενημέρωσης για τα, για τα μέτρα που αναλαμβάνονται. Η Επιτροπή αναλαμβάνει τον έλεγχο των συστημάτων όπως τα προβλέπουν τα κράτη-μέλη. Επίσης η επιβολή του προγράμματος θα είναι υποχρεωτική και για αυτό το σκοπό η Επιτροπή θα μπορεί σε μόνιμη βάση να ελέγχει τον τρόπο κατά τον οποίο τα κράτη-μέλη φέρνουν εις πέρας αυτές τις υποχρεώσεις. Η οδηγία καλύπτει όλα τα αναλωμένα καύσιμα και τα ραδιενεργά απόβλητα ε, που χρησιμοποιούνται για πολιτικούς σκοπούς. Μιλάμε για προϊόντα που δεν χρησιμοποιούνται στα εργοστάσια παραγωγής ε, πυρηνικής ενέργειας, ούτε είναι αποτέλεσμα απευθείας εξόριξης. Εδώ θέλουμε να αποφύγουμε την επικάλυψη και με άλλες οδηγίες. Λόγω χάρη οδηγία που αφορά τα διενεργά απόβλητα από, από εξόριξη. Εκεί υπάρχει ειδική νομοθετική πράξη. Τώρα να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένη. Η οδηγία αυτή προβλέπει και αρμόδια ρυθμιστική αρχή στον τομέα αυτό. Επιπλέον, ορίζει τις ευθύνες του υπεύθυνου της ε, παραγωγής προβλέπονται μέτρα για την εκπαίδευση και την κατάρτιση με ειδικά άρθρα επίσης ειδικά άρθρα για την διαφάνεια όπου προβλέπεται για τα κάτι μέλη υποχρέωση να ετοιμάσουν ειδικό πρόγραμμα. Επίσης προβλέπεται η, η εξέταση της ασφάλειας, η αξιολόγηση της ασφάλειας με ειδικά συστήματα και διαδικασίες και επίσης υπάρχει απέτηση για επαρκείς ε, πόρους σηματοδότησης. Η δική μου πρώτη αποτίμηση της οδηγίας πιστεύω ότι είναι πολύ θετικό να έχουμε αυτή την οδηγία την πρόταση οδηγία επιτάπητο. Νομίζω ότι η προετοιμασία τη είναι αρκετά ικανοποιητική, λαμβάνοντα υπόψη τι είναι γενικώ αποδεκτό σε αυτή τη χρονική περίοδο. Παρόλα αυτά, σε ορισμένα σημεία θα ήθελα η οδηγία να είναι πιο έντονη στις ε, υποχρεώσει που προβλέπει, ισχυρότερη. σε κάποια σημεία είναι λίγο αδύναμη, σε άλλα σημεία επίση βρίσκω ότι οι απαιτήσει παρά είναι αυστηρέ. Δεδομένη τη κατάσταση όπω σήμερα έχει διαμορφωθεί βεβαίω. Επίση, να προτείνω κάποιους επιπλέον ορισμούς ε, σε σχέση με που θεωρώ ότι λείπουν. Για τον ορισμό των ενεργών αποβλήτων, φαντάζομαι ότι αυτός μπορεί να συζητηθεί. Ε, και είναι και απαραίτητη μια τέτοια συζήτηση. Πρέπει να δούμε κατά πόσον είναι αντιστρέψιμη όλη η διαδικασία. Προς τον ορισμό αυτό. Κάτι ακόμη. Η οδηγία μιλάει για επαρκή ανθρώπινους πόρους, εκπαίδευση και κατάρτιση. Δεν υπάρχουν ειδικέ απαιτήσει για την έρευνα και τι ε, ενέργειε ε, δράση ανάπτυξη. Η οδηγία επίσης ορίζει ότι πρέπει να προσφέρεται επαρκής γνώση για τη διαχείριση των ερευνητικών αποβλήτων και των αναλωμένων καυσίμων αλλά δεν κάνει λόγο για την παρακολούθηση, για monitoring. Θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει ισορροπία σε όλα τα τμήματα του κειμένου μεταξύ τους, άρα να κοιτάξουμε πώς θα αναδιατυπώσουμε κάποια σημεία των άρθρων. Κάποια άρθρα περισσότερο αρμόζουν στην οδηγία για την πυρηνική ασφάλεια παρά σε αυτήν. Λαμβάνοντα υπόψη το έργο του Ευρωκοινοβουλίου στο παρελθόν για τους σηματοδοτικούς πόρους και υπό το φως όλων αυτών των στοιχείων, νομίζω ότι τελικά η οδηγία είναι αρκετά αδύναμη. Όμως πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές στην προσέγγιση μας. Δεν θα πρέπει να υποβάλουμε ένα κατάλογο με το τι θα επιθυμούσαμε να συμβεί, αλλά να δούμε τι μπορεί να γίνει αποδεκτό σε αυτή τη χρονική φάση και τι θα είναι ρεαλιστικό στην προσέγγιση μας. Ως προς τη διαφάνεια. Η Επιτροπή μελετά το πώς θα μπορέσει να συμπεριλάβει στην όλη διαδικασία και το κοινό, τους πολίτες. Εμείς διαρωτόμαστε κατά πόσον διαφάνεια σημαίνει κάτι παραπάνω από αυτό. Μήπως πρέπει να συμπεριλάβουμε ορισμό για τη συνεργασία και τη συμμετοχή του κοινού βάσει της ε, σύμβασης του άρχους. Θα πρέπει να κοιτάξουμε να λαμβάνονται και αποφάσεις και να αποδοθούν αρμοδιότητες ώστε να λαμβάνονται αποφάσεις. Η οδηγία, αυτή, ε, η οδηγία εδώ δεν είναι σαφής. Θα αναποθέτω λεφτά στην ε, κρίση των κρατών μελών. Τώρα, για τις συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών. Τέτοιες συμφωνίες ήδη υπάρχουν, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και δεν πρέπει να συμπεριφερόμαστε σαν να τις αγνοούμε. Κάποιες περιφερειακές πρωτοβουλίες επίσης προτείνονται. Εδώ θα πρέπει να σχεδιάσουμε κάποιο πλαίσιο για αυτές τις περιφερειακές πρωτοβουλίες. Να αποφύγουμε να γίνουν αυτές οι πρωτοβουλίες πρόσχημα ώστε τα κράτη-μέλη να αναβάλουν τη λήψη αποφάσεων στο μέλλον. Επίσης, πρέπει να σκεφτούμε την απέτηση για πλήρη απαγόρευση εξαγωγής ραδιενεργών αποβλήτων. Υπάρχουν κάποιες δράσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, προς αυτή την κατεύθυνση. Κάποια πράγματα γίνονται αποδεκτά, όπως η διαχείριση για τους αντιδραστήρες, στην περίπτωση των αντιδραστήρων. Και κάτι ακόμη. Πώς η ομάδα ENSREC μπορεί να αναλάβει εδώ ε, ευθύνε για, για τέτοιε δραστηριότητε. Μιλάω για την ε, ομάδα των Ευρωπαίων ε, Ρυθμιστών Πυρηνική ενέργεια. Αυτές ήταν οι μου για την οδηγία. Είμαι πρόθυμο να συνεργαστώ με όλους σα. και θα λάβω σοβαρά υπόψη και τι ε, δικέ σα προτάσει, τι τροπολογίε σα για να βελτιωθεί η έκθεση. Επίση, να απευθύνω έκκληση προ του εκπροσώπου του Συμβουλίου. Πώ έχετε σκεφτεί εσεί τη συνεργασία μαζί μα. Θα ήθελα κάποια εγγύηση από την πλευρά σα ότι όσα κάνουμε δεν θα είναι ει ότι το Συμβούλιο θα λάβει υπόψη όσα εδώ εγκρίνουμε σε επίπεδο επιτροπή μα και στην Ολομέλεια βεβαίω. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Παρακαλώ να αρχίσουμε τώρα τη συζήτηση. Ζήτησαν μερικοί ήδη το λόγο, αλλά θα πρέπει να οργανώσουμε το χρόνο μας έτσι, τους, ώστε να μπορέσουμε να πραγματευτούμε και το σημείο 11 της ημερήσιας διάταξης πριν, πριν από τις ψηφοφορίες. Ο κύριος Μεζαρός, Μεζάρος έχει το λόγο πρώτος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Γιόρνταν Σιζέλ για την, την εισηγήτρια για την ε, παρουσίασή της. Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό θέμα και χαίρομαι που τώρα συζητούμε μια οδηγία η οποία μπορεί να παράσχει λύση. Εδώ θίγονται όλες οι χώρες και στη χώρα μου, στη Σλοβακία, 70% της ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται από πυρηνική ενέργεια. Η θα πρέπει βεβαίως από ό,τι κατάλαβα να καταλήξουμε σε κάποια συμβαστική λύση μεταξύ πολύ αυστηρών και χαλαρότερων διατάξεων. Δεν θα πρέπει να είμαστε υπερβολικά αυστηροί, δεν θα πρέπει η πυρηνική ενέργεια να είναι υπερβολικά ακριβή. Αλλά ε, δυστυχώς παράγονται ραδιενεργά απόβλητα, ραδιοϊσότοπα και όχι μόνο στους αντιδραστήρες. Ε, υπάρχουν διάφορες ε, δυνατότητες βέβαια εδώ υπάρχει ε, η δυνατότητα ανακύκλωσης αυτών των ραδιοεισοτόπων υπάρχει και βεβαίως η δυνατότητα της α, απομάκρυνσης. Ε, έχουμε τρεις κατηγορίες τέτοιου είδους αποβλήτων και τρεις μεθόδους άρα διαχείρισης των αποβλήτων αυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε η συγγήτρια εδώ, ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε με το Συμβούλιο και να ε, πιέσουμε αν είναι δυνατόν το Συμβούλιο να λάβει υπόψη τις και τις δικές μας συστάσεις. Και είναι πολύ σημαντικό επίσης και αυτό που είπε η συγγήτρια για τις εξαγωγές αποβλήτων. Είναι πολύ σημαντικό να μην συμφωνήσουμε να τα απόβλητα τα οποία δημιουργούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εξάγονται και να απομακρύνονται στο εξωτερικό. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και πρέπει να, να το προσέξουμε. Η οδηγία επίσης δεν αναφέρεται καθόλου στην ασφάλεια των μεταφορών των αποβλήτων αυτών. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Και δύο λόγια πριν κλείσω. Ε, πολλά χρόνια, εδώ και πολλά χρόνια και σε πολλές χώρες μέλη υπάρχει ένα κίνημα ενάντια στην πυρηνική ενέργεια. Ε, η παρόλο που οι ειδικοί ε, μιλούν για μεγάλες αλλαγές στην πυρηνική ενέργεια και για αύξηση του επίπεδου ασφαλείας, τους αντιδραστήρες κτλ. Καλό θα ήταν λοιπόν να υπάρχει και κάτι μέσα στην οδηγία που να προωθεί την έρευνα ιδιαίτερα σε σχέση με θέματα ασφάλειας και την ε, κατάρτιση για την πυρηνική ενέργεια. Αυτά από πλευράς μου. Ε, Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Ε, ναι, είναι δική σου σειρά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα πρέπει να σας πω ότι προσωπικά είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος το ότι επιτέλους συζητούμε αυτό το σημαντικό θέμα όσον αφορά ε, αυτή τη, διαχείριση αυτών των ε, ουσιών, αποβλήτων κλπ. σε κάποιο ενωσιακό, συντονισμένο το σε επίπεδο και τελικά όπως όλοι γνωρίζουμε και πρέπει όμως να το επενθυμίζουμε, πρόκειται για τη δεύτερη προσπάθεια που καταβάλαμε ε, από τότε που ξεκίνησαν το 2004 οι σχετικές διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο, τότε είχαμε τη σχετική οδηγία δηλαδή για τα απόβλητα. Εγώ θυμάμαι ότι ήμουν ο εισηγητής επ' αυτού, όμως δυστυχώς δεν κατέστη δυνατόν να αποσπάσουμε το πρόβλημα το οποίο θέλαμε τότε. Ε, σήμερα τα πράγματα έχουν ε, αλλάξει. Η οδηγία για την ασφάλεια ήδη τον Ιούνιο ε, ε, είχε περάσει τον Ιούνιο του 2009 επομένως είπαμε και τώρα μπαίνουμε σε μια καινούργια εποχή, σε μια εποχή ε, που ξεκίνησε όπως είπαμε το 2003-2004 η πρώτη φάση και σήμερα μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε μια εποχή αναγέννησης για ε, τη διαχείριση των πυρηνικών, οπότε έχει διαμορφωθεί μια ευρεία συνένεση στην ε, διεθνή επιστημονική κοινότητα ε, όσον αφορά το ότι η, η, η διαχείριση με ταφή γεωλογική σε μεγάλο βάθος είναι η πιο δόκιμη λύση και επομένως θεωρούμε ότι τώρα μπορούμε να έχουμε μια στέρεα βάση όσον αφορά κάποια συμπράσματα που μπορούμε να εξαγάγουμε. Τώρα όσον αφορά το περιεχόμενο της οδηγίας, εγώ συμφωνώ 100% με τις απόψεις, με τις ε, σκέψεις ε, της ε, Ρωμάνα Τζόρνταν και νομίζω επομένω ότι είναι πάρα πολύ σωστή, συνεπή αυτή η οδηγία, οπότε και συμφωνώ και με αυτή τη φόρμουλα των δύο φάσεων που υπηρετεί τη συνέχιση τη αρχική προσπάθεια για να έχουμε έτσι αυτή την, ε, ε, τον συμβασμό μεταξύ των εθνικών προσπαθειών, εθνικών προγραμμάτων και από την άλλη μεριά αυτού το οποίο χρειάζεται τόσο πολύ, δηλαδή να υπάρχει ένας συντονισμός ευρωπαϊκός ακόμα και με το να έχουμε ε, την δυνατότητα να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν το εθνικό πρόγραμμα τελικά ε, αποδειχθεί ασυνεπές, ανεπαρκές σε αυτό το άρθρο. Επίσης όσον αφορά την αρχή επί των ε, χρηματοοικονομικών συμφωνώ στο άρθρο 10. Εκεί νομίζω ότι εξυπηρετείται ο βασικός στόχο, ότι δηλαδή τα χρήματα θα πρέπει να εκταμιεύονται να είναι διαθέσιμα όταν χρειάζονται. Κατά τα λοιπά, η έκθεση είναι πάρα πολύ καλά διαδρομένη, καλύπτει τα θέματα τα βασικότερα. Βέβαια θα πρέπει να χτενίσουμε κάποια σημεία, δηλαδή τον ορισμό του ρεδινεργού αποβλήτου, τις εξαγωγικές, ε, τους περιορισμούς τέλο πάντων ε, και τα σχετικά με την ασφάλεια. Πάντως ε, νομίζω ότι εν γέννη μπορούμε να τη βελτιώσουμε την οδηγία. Οπότε για άλλη μια φορά συγχαρητήρια στην Ρωμάνα και μπορεί οπωσδήποτε να υπολογίζει ή στην αμέριστη συμπαράστασή μας. Ευχαριστώ εγώ ευχαριστώ. Είσαι συνάδελφος Thank you. Um, ευχαριστώ. Πρώτα πρώτα, λέει κύριε Χολ, να ευχαριστήσω την ε, εισηγήτρια για το ότι προέβη σε όλες αυτές τις διαβουλεύσεις με τους χιώδες εισηγητές. Αυτό είναι θετικό, είναι βήματα προόδου και θα έχουμε και ευκαιρίες να τα πούμε. Επίσης σας ευχαριστούμε διότι η ανάλυση που κάνατε ήταν πάρα πολύ ε, ενδελεχής όσον αφορά μια σειρά ζητημάτων τα οποία οπωσδήποτε και είναι πάρα πολύ σημαντικά για το θέμα μας. Ε, επίσης μας ικανοποίησε πάρα πολύ το ότι αναφέρατε ε, την πτυχή της ενιαίας αγοράς διότι αυτό ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη δυναμία στο παρελθόν διότι επανειλημμένα στο παρελθόν ε, το, το, κόστος του να κλείσει ένα σταθμός, του να διαχειριστούν αυτά τα, διαχειριστούν αυτά τα απόβλητα ε, θεωρήθηκε ότι δεν υποστηρίζεται οικονομικά όπως θα έπρεπε και επομένως ε, τελικά ε, πρόκειται για πολυδάπανη εργασία αλλά δεν αντικατοριζόταν αυτό στο κόστος του ηλεκτρισμού το οποίο, ο οποίος ε, είχε παραχθεί με ε, την πυρηνική ενέργεια. Πάντως, εγώ έχω κάποιες, κάποιους προβληματισμούς πάρα πολύ σοβαρούς όσον αφορά τα, τα, τα επιχειρήματα τα οποία ε, βρίσκονται πίσω από την πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. επιτροπης Επιτροπής. Συγκεκριμένα, πρώτα-πρώτα λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λέει ότι υπάρχει μια ευρεία συνένεση, γενική συνένεση, για το ότι η, η ταφή σε μεγάλο βάθος είναι η πιο δόκιμη λύση για την ενεργά απόβλητα. Όμως, ε, εγώ τώρα μου έρχονται στο μυαλό οι ηλικιωμένες χωρών που λένε ότι αυτό είναι ε, ο άγνωστος χ. Λέει εδώ πέρα η Κομισιόν ότι υπάρχει ευρεία συνένεση, αλλά δεν παρέχει καμία τεκμηρίωση ε, όσον αφορά δηλαδή το με ποια έρευνα προέκυψε αυτό. Επομένως, θα βοηθούσε πάρα πολύ ε, αν αυτού του τη, μυστηριώδη τεκμηρίωση μας την παρέσχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να δούμε ακριβώς ποια μπορεί να είναι η μακρόπνοη λύση, γιατί η εμπειρία μας λέει ότι η διαχείριση ρεδινεργών αποβλήτων είναι πολύ περίπλοκο θέμα. Και μιλούμε τώρα για μεσοπρόθεσμη αποθήκευση. Στο Ηνωμένο Βασίλειο είχαμε προσέξει ιδιαίτερος για να εξασφαλίσουμε το τι θα γίνει εάν έχουμε κάποιο σεισμό σε σχέση με τον χώρο αποθήκευσης των αποβλήτων. Ούτω ώστε το κοντέν, ο περιέκτης αυτών των αποβλήτων να μην υποστεί κάποια ζημιά. Όμως από την μεριά υπάρχει κόπωση του υλικού του μετάλλου και τι θα γίνει αν έχουμε ένα σωρό ραδιενεργό υλικό το οποίο θα διαρρεύσει. 83 ξέρω εγώ κυβικά ε, ας πούμε με κάποιο είδου γυαλί και το άλλο πρόβλημα το οποίο βγαίνει και από την πρόταση της Κομισιόν είναι το ότι ενδεχομένως υπάρχει εδώ σύγκρουση μεταξύ αυτού που τεχνοκρατικά είναι το πιο προτιμητέο και από την μεριά αυτό το οποίο ε, προτιμάει ο κόσμος. Γι' αυτό και ίσως θα πρέπει να γίνει διαβουλεύση και με τον κόσμο για το τι θα προτιμήσουμε. Οπότε έχουμε τώρα αυτού του είδους τις πυρηνικές εγκαταστάσεις ή έχουμε εκεί το χώρο αποθήκευσης και ο σχετικός χώρος είναι αποδεκτός από τον, από, από τον κόσμο. Ενώ από την άλλη μεριά λέμε το ότι να είναι κάπου σε ένα πάρκο βαθιά θαμμένα είναι αυτό το οποίο οι τεχνοκράτες προτιμούν και να δούμε τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφού μελετήσει τις εκθέσεις των κρατών μελών της, αναφορές όλα αυτά και πώς θα, τι, τι θα προτιμήσουν, θα προτιμήσουν αυτό που τεχνικά είναι προτιμητέο ή αυτό που προτιμάει ο κόσμος. Έχουμε μόνο εδώ κάποια περίπλοκα ζητήματα τα οποία δεν νομίζω ότι τα απαντά, τα επιλύει τέλος πάντων το κείμενο της Κομισιόν. Κύριε Χάρμς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω πρώτα-πρώτα ότι η συζήτηση αυτή θα πρέπει να γίνει με διαφορετικό τρόπο από, από ό,τι έγινε η συζήτηση ας πούμε για την ατομική πυρηνική ενέργεια. Δεν μπορούμε να είμαστε υπέρ ή κατά. Τα απόβλητα δημιουργούνται και πρέπει οπωσδήποτε να απομακρυνθούν με κάποιο τρόπο. Άρα λύση πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί. Σε καμιά από τις χώρες που αυτή τη στιγμή έχουν πυρηνικούς αντιδραστήρες και παράγουν πυρηνική ενέργεια δεν υπάρχει τελικός χώρος αποθήκευσης αυτών των αποβλήτων και αυτό ε, δημιουργεί πρόβλημα μπορεί να γίνεται μια κάποια διαχείριση αλλά δεν υπάρχει χώρος τελικής ε, διατήρησης, αν θέλετε, φύλαξης αυτών των αποβλήτων στη δική μου τη χώρα, στη, ιδιαίτερα στην κάτω Σαξονία που είναι η δική μου η περιοχή, ε, έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες και ε, ε, ε επελέχθη ένα οριχείο ε, άλατος στο οποίο γινόταν η ταφή αυτών των αποβλήτων ε, εδώ και, και πολλά χρόνια. Αυτή τη στιγμή όμως η κατάσταση σε αυτή την περιοχή ε, η κατάσταση έχει γίνει τραγική. Δεν υπάρχουν μέθοδοι να εξασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχουν επιπτώσεις. 30 χρόνια μετά την αναρχική η χρήση αυτού του ορυχείου αν θέλετε ως αποθήκης αυτών των αποβλήτων ε, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε με τα βαρέλια στα οποία τα οποία είναι σφραγισμένα και τα λοιπά και στα οποία μπαίναν αυτά τα απόβλητα δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε ή δημιουργούν προβλήματα όπως μας έχουν διαβεβαιώσει οι γεωλόγοι η κατάσταση είναι τραγική. Αυτή η περίπτωση ήταν πρώτη χρησιμοποιήθηκε σαν μοντέλο στη χώρα μου για τελή την τελική αποθήκευση αυτών των αποβλήτων και τώρα βλέπουμε τα χάλια στα οποία έχουμε φτάσει η Ευρατόμ πρόκρινε αυτού του είδους την φύλαξη ε, δεν είναι λοιπόν καθόλου σίγουρο ότι η ταφή ακόμη και αν είναι σε βάθος 700 μέτρα όπως αυτό το συγκεκριμένο ορυχείο είναι λύση πρέπει να προσέξουμε Χτες Χτε ο, ο Επίτροπος ε, στην αρχή της ανάληψης της θητείας του είχε πει ότι το κόστος είναι... Δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη εδώ καθόλου, διότι η φύλαξη, αποθήκευση ραδιενεργών αποβλήτων είναι τόσο σημαντικό θέμα και μπορεί να επηρεάσει τόσο πολύ μελλοντικέ γενιές που δεν θα πρέπει να μας ενδιαφέρει το κόστος. Θα πρέπει να, να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση. Συμφωνώ λοιπόν με αυτό που είπε ο Επίτροπος και γι' αυτό έχω διάφορα ερωτηματικά και για τούτη εδώ την οδηγία. Δεν μπορώ να καταλάβω, ε, παραδείγματος χάρη γιατί αποκλείονται από εδώ τα προϊόντα ουρανίου. Γιατί δεν αναφέρεται εδώ καθόλου η στρατιωτική χρήση. Τα στρατιωτικά απόβλητα δηλαδή θα πάνε τελείως χωριστά ε, από τα άλλα απόβλητα. Αν έχουμε ένα και δύο και τρία μέρη όπου αποθηκεύονται απόβλητα σε μια χώρα, τότε διπλασιάζουμε, τριπλασιάζουμε το ρίσκο, τους κινδύνους που υπάρχουν από τους χώρους αυτούς, τα φύση ή τέλο πάντων φύλαξης. Υπάρχουν λοιπόν πολλά ερωτηματικά εδώ και πραγματικά Υπάρχουν ας πούμε εκπομπές, υπάρχουν και άλλα απόβλητα τα οποία δεν καλύπτονται από την οδηγία αυτή. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Αν θέλουμε πάντως να φτιάξουμε μία οδηγία για την διαρκή φύλαξη αυτών των αποβλήτων δεν μπορούμε να αποκλείουμε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Επίσης νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε το θέμα της συμπερίληψης, ε, της συμμετοχής εδώ των πολιτών, του κοινού όπως ελέγχθη. Υπάρχουν κανόνες της Ευρατόμ, ε, που επιτρέπουν τη συμμετοχή αν θέλετε αλλά πέραν αυτών το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οποιοδήποτε κοινοβούλιο θα έπρεπε να έχει τη δυνατότητα να προσελκύσει το, το κοινό και να εμπλέξει το κοινό συζήτηση τέτοιου είδου θεμάτων το European Nuclear Energy Forum παραδείγματο χάρη θα μπορούσε να εμπλέξει το κοινό και η Κομισιόν θα έπρεπε να συνεργαστεί με αυτό. Α, και η πυρηνική οικονομία, αν θέλετε, η κλάδο κοινωνικής οικονομία που σχετίζεται με την πυρηνική ενέργεια ζητεί, αν δεν κάνω λάθο, ε, την συμμετοχή των πολιτών. Και ε, ε, γι' αυτό σας λέω ότι λείπουν κάποια πράγματα από την ε, ε, οδηγία για την ε, φύλαξη, για την αποθήκευση ε, και για την απομάκρυνση την τελική των αποβλήτων. Εγώ ως Γερμανίδα σας λέω ότι δεν μπορούν να πάρθουν αποφάσεις χωρίς η συμμετοχή του κοινού, χωρίς σοβαρές συζητήσεις με το κοινό. Γιατί υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα τα οποία πορέουν από τις έρευνες των τελευταίων δεκαετιών και που πρέπει να ε, επιληθούν. Όπως είπε και η συνάδελφος Χολ υπάρχουν πράγματα που σχετίζονται παραδείγματο χάρη με το κατά πόσον είναι αντιστρέψιμες κάποιες δράσεις τις οποίες αναλαμβάνουμε. δηλαδή τώρα αποφασίσουμε να φυλάξουμε τα απόβλητα αυτά με τον αλφα τρόπο μπορούμε να αντιστρέψουμε την κατάσταση στο μέλλον. Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα αυτό ειδικά στη βιομηχανοποιημένη Ευρώπη, Δυτική Ευρώπη αυτή τη στιγμή τα προβλήματα είναι τεράστια. Ε, πολύ λίγες χώρες στον κόσμο έχουν τόσα προβλήματα. Γι' αυτό πραγματικά παρακαλώ όλα αυτά τα θεμελιώδη ερωτήματα τα οποία ακόμη δεν έχουν καλυφθεί από την οδηγία να τα α, συζητήσουμε τουλάχιστον εμείς. Βλέπω ότι υπάρχει μια κάποια ανυπομονησία από πλευρά ορισμένων και από τη δική σας πλευρά κύριε Πρόεδρε, αλλά θεωρώ ότι είναι τόσο μεγάλη σημασία στα θέματα αυτά που θα πρέπει να κάνουμε υπομονή ε, δεν πρόκειται για δευτερεύον θέμα, πρόκειται για τα πάρα πολύ ε, σημαντικό θέμα. Πρόεδρος, αγαπητή κυρία Χάμσε, έχω υπομονή, είμαι υπομονετικός άνθρωπος και καταλαβαίνω πόσο σημαντικά είναι τα θέματα αυτά. Απ' την άλλη μεριά όμως, εγώ ως πρόεδρος είμαι υποχρεωμένος να ε, διαχειριστώ και το χρόνο, διότι αν συνεχίσετε συνεχίσουν όλοι να μιλούν τόσο πολύ όσο μιλήσατε εσείς, κάποιοι άλλοι δεν θα μπορέσουν να πάρουν το λόγο. Γι' αυτό κάπως εκνευρίστηκα αν θέλετε και έδειξα μια κάποια ανυπομονησία τίποτε παραπάνω λοιπόν η κυρία Χέρτσοκ έχει τώρα το λόγο αν δεν έχω κανένα πρόβλημα μπορούμε να μείνουμε μέχρι το βράδυ εδώ έτσι αλλά δεν θα υπάρχει κανείς στην αίθουσα η κυρία Χέρτσοκ Καλημέρα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Άρχισα λιγάκι, διότι βρισκόμουν και σε άλλη επιτροπή. Ως ε, σκιώδης για τους σωλιστές, θέλω να συμμετάσχω προφανώς. Να ευχαριστήσω λοιπόν ιδιαίτερα την συγκεκριά μας και τους σκιώδης. Ε, νομίζω ότι ε, ήταν πολύ επιτυχη η συνεργασία μας ως τώρα, μάλιστα ήδη από τις πρώτες συναντήσεις μας. Συζητήσαμε και συμφωνήσαμε για το χρονοδιάγραμμα, μπορούμε να συμφωνήσουμε γι' αυτό. Θέλω να, να αναφέρω ότι η Ουγγρική Προεδρία με ιδιαίτερη ικανοποίηση θα ολοκληρώσει την εξέταση του θέματος αυτό, όπως ακούσαμε χθε από τον Υπουργό στο εξάμεινό τη και πιστεύω ότι παρόλο πρέπει να συζητήσουμε όλα τα σημαντικά ζητήματα με όσο το δυνατόν πιο προσεκτικό τρόπο, παρόλα αυτά δεν πρέπει να ξεχνάμε τι ημερομηνίε μπορεί να ακολουθήσει και το Συμβούλιο, κυρίω επειδή το Ευρωκοινοβούλιο εδώ έχει μόνον συμβουλευτικό ρόλο. Η οδηγία αυτή είναι μέρος και βασίζεται μάλλον στη συνθήκη Ευρατόμ. Τώρα, η συνθήκη Ευρατόμ έχει το βασικό πλεονέκτημα ότι ο μόνος τρόπος να επιτευχθεί πρόοδος να επιτελεστεί πρόοδο είναι να συμφωνήσουν τα 27 κράτη-μέλη. Το Ευρωκοινοβούλιο εδώ έχει απλώ συμβουλευτικό ρόλο, όπω είπαμε. Όμω κάποιες συζητήσεις, κάποια σημεία που αφορούν τα ραδιενεργά μπορεί να βασιστούν στη συνθήκη της Λισαβόνας, οπότε εκεί το Κοινοβούλιο μπορεί να έχει ενισχυμένο ρόλο να διαδραματίσει. Πάντως είναι πολύ σημαντικό η Επιτροπή Ήτρε να το λάβει το θέμα αυτό υπόψη πολύ σοβαρά. Οι σκιώδεις εισηγητές ούτως ή άλλως σας διαβεβαιώ, το λαμβάνουν σοβαρά, θα εξετάσουν τα ζητήματα με ιδιαίτερη προσοχή και θέλουμε να έχουμε ευκαιρίε να συζητήσουμε ώστε και το κοινό να γνωρίζει τι κάνουμε εδώ να προβληθεί το έργο μας. Νομίζω ότι το βασικό ζήτημα που πρέπει να μας απασχολήσει και να αποφασίσουμε σε σχέση με την οδηγία είναι τι είναι πιο σημαντικό. Έχουμε υψηλέ φιλοδοξίες Το θέμα όμω είναι μήπω κάποιο τελευταία στιγμή αλλάξει γνώμη, αλλάξει τη συμφωνία και δεν θέλει να ακολουθήσει. Οπότε στο τέλο θα καταλήξουμε στο μηδέν. Ή να πηγαίνουμε βήμα προ βήμα, ε, ίσω πιο αργά, αλλά να συμφωνούμε όλοι μεταξύ μα. Οπότε στα εμπόδια, στι δυσκολίε όπου δεν θα μπορούμε να συμφωνήσουμε, ε, με μελλοντικέ διαπραγματεύσει να μπορούμε να επιτελέσουμε κάποια πρόοδο. Εγώ νομίζω ότι η δεύτερη προσέγγιση είναι καλύτερη. Δηλαδή, ό,τι πρέπει να φύγει από την οδηγία αυτή αργά ή γρήγορα, θα είναι ένα τίμημα που θα καταβάλουμε προκειμένου να επετελεστεί όμως ένα βήμα πρόοδου. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας ευθύς εξ αρχής. Επίσης, ως προς τη γενική μας προσέγγιση, ε, μάλλον μετά τη γενική μας προσέγγιση, να κάνω κάποια συγκεκριμένα σχόλια και ερωτήματα. Η ευθύνη των κρατών μελών πρέπει να παραμείνει, σε αυτό συμφωνούμε όλοι, όμω από την άλλη βλέπουμε ότι οικονομική κλίμακα, ούτε η κλίμακα πραγματική υλοποίηση των μέτρων αυτών είναι δυνατόν να έρθει πέρα από τα κράτη-μέλη και μόνον. Στι ΗΠΑ, λόγω χάρη, αναζητούν μία τελική λύση, ένα τελικό σημείο. Ή θα αφήσουμε λοιπόν τα κράτη-μέλη να βρουν ξεχωριστέ λύσει, ή θα πρέπει να άρουμε του πολιτικού φραγμού και του φραγμού τη αγορά αυτούς που υπάρχουν σήμερα για να δούμε σε ευρύτερη κλίμακα τι λύση μπορεί να δοθεί συνολικά. Τι μπορεί να γίνει και τι μπορεί να δεχτεί βεβαίω και το κοινό, οι πολίτες. Επίσης θα πρέπει να επεξεργαστούμε λίγο ε, τους ορισμούς των αδιενεργών αποβλήτων και των ανελωμένων καυσίμων, διότι κάποιες φορές σχετίζονται με το επόμενο σημείο που θέλω να θίξω. Δηλαδή, να σκεφτούμε τι εννοούμε εξαγωγές και τι εννοούμε χώρα προέλευσης για τα απόβλητα. Εννοούμε χώρα προέλευσης εκεί όπου παράχθηκε ενέργεια ή υπήρξε οποιαδήποτε άλλη χρήση της ή εκεί που υπήρχε επεξεργασία. Ε, να ορισμένες από τις υποθέσεις. Ε, επίσης, νομίζω το στοιχείο αυτό θα απασχολήσει ιδιαίτερω και το Συμβούλιο και θέλουμε να υποστήλουμε ένα μήνυμα εδώ και από το Ευρωκοινοβούλιο. Δηλαδή, να συμφωνήσουμε εκεί όπου μπορεί να υπάρχει συμφωνία και να προχωρούμε. Ε, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί λοιπόν, γιατί εδώ υπάρχει υπάρχουν διασυνδέσεις και με την οδηγία για την ασφάλεια των, ε, την, της ασφάλειας. Θα πρέπει λοιπόν να εξεύρουμε μία λύση ώστε να συμβαδίζουν οι δύο οδηγίες. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε εδώ είναι ό,τι συζητήσουμε περί ασφάλειας να μην ξεπερνά τα όρια τη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων. Διότι ο οδηγία αυτό το θέμα ακριβώ αφορά. Δεν θέλουμε να επιλύσουμε όλα τα ζητήματα ασφάλεια που έχουν να κάνουν με την πυρηνική βιομηχανία εδώ. Δεν νομίζουμε ότι είναι και κατάλληλος, κατάλληλη ευκαιρία. Ε, θα πρέπει να γίνει ξεχωριστή συζήτηση και πιστεύουμε για τα ζητήματα που μα αφορούν να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε. Τέλο, για τη διαφάνεια και την ενημέρωση του κοινού. Νομίζω ότι αν Υπάρχει ένα βιομηχανικό κλάδο στην Ευρώπη που κατάλαβε πόσο σημαντική είναι η ενημέρωση του κοινού, είναι ακριβώ η πυρηνική βιομηχανία, η βιομηχανία τη ραδιενέργεια. Είδαμε με τι πετρελαϊκέ εταιρείε πόσο πίσω είναι σε σχέση με την ε, βιομηχανία των πυρηνικών. Θα πρέπει λοιπόν ε, να. τη πυρηνική ενέργεια. Θα πρέπει να το έχουμε αυτό υπόψη. Το κοινό πρέπει να ενημερώνεται, πρέπει να συμμετέχει. Αυτός είναι ο τρόπος να προχωρήσουμε και ίσως αυτό είναι κάτι παραπάνω από την απλή διαφάνεια. Νομίζω όμως ότι μεταξύ μας θα καταφέρουμε να εξεύρουμε μια κατάλληλη λύση και ελπίζω να παραμένουμε πιστοί και στο χρονοδιάγραμμα. Πρόεδρε, το Συμβούλιο δεν θα προχωρήσει έτσι καλλιώς χωρίς τα δικά μας πορίσματα από τις διαβουλεύσεις μας. Θα συνεργαστούμε λοιπόν με τον εισηγητή και θα, με όλους σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά σύντομα όμως. Ε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, όντως θα είμαι σύντομος. Πρώτα-πρώτα πιστεύω κι εγώ μετά τις παρεμβάσεις και της εισηγήτριας και των σκιωδών εισηγητών ότι έγινε σαφές ότι εδώ ε, θίγονται αν θέλετε ε, και οι 27 χώρες. Όλες οι χώρες παράγουν ραδιενεργά απόβλητα είτε έχουν αντιδραστήρες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είτε όχι διότι υπάρχουν και η έρευνα και τα νοσοκομεία κτλ τα δεν χάρηκα ιδιαίτερα από την παρέμβαση της κυρίας Χάμς η οποία λέει ε, δεν ε, είναι και χάρηκα ιδιαίτερα, με συγχωρείτε, για την παρέμβαση της κυρίας Χάμς που είπε ακριβώς το δεο δεν πρόκειται για ένα υπέρ ή ένα κατά, πρέπει να επιληθούν τεχνικά θέμ και τεχνικά θέματα. Εμείς από πλευρά Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα είμαστε πρόθυμοι να εξετάσουμε απόψεις ε, να ψάξουμε επιστημονικά δεδομένα και να βρούμε μια επιστημονική συνένεση. Αλλά επιστημονική συνένεση δεν είναι το ίδιο με κοινωνική συνένεση. Η διαφάνεια και η συμμετοχή των πολιτών είναι άλλο πράγμα από την επιστημονική συνένεση. Το φινλανδικό και σουηδικό παράδειγμα έδειξε ότι βεβαίω ορισμένε αποφάσει δεν μπορούν να παρθούν και ορισμένα πράγματα δεν μπορούν να προχωρήσουν αν δεν στηριχθούν από την τοπική κοινωνία. Αλλά καταλάβετε κιόλας ότι ούτε η Κομισιόν, ούτε το Συμβούλιο, ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν τη νομική βάση αυτή τη στιγμή, εφόσον μιλάμε για την συνθήκη Ευρω... Ευρατόμ, να προσθέσουν θέματα εδώ, όπως παραδείγματο χάρη στρατιωτικές χρήσεις κτλ. Δεν είμαστε σε θέση να υποβάλουμε εμείς σαν Κομισιόν, δεν δεν, έχουμε αυτό το δικαίωμα να υποβάλουμε προ, προτάσεις για τις ε, τα στρατιωτικά απόβλητα. Το θέμα των εξαγωγών, το θέμα της ασφάλειας είναι θέματα που μπορούν να συζητηθούν και υπάρχουν πολλές δυνατότητες αλλά μια και δεν υπάρχει πολύς χρόνος όπως είπε και ο πρόεδρος ε, δεν ε, θα συνεχίσω θα πω απλώς ότι η η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ανα πάσα στιγμή στη διάθεσή σας, στη διάθεση της συγγήτριας, των σκιωδών εισηγητών και θέλουμε να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Θέλεις Ρωμάνα και πάλι το λόγο. Δύο λόγια μόνο. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τα σχόλια τους. Είναι πολλά τα προβλήματα, πολλές οι δυσκολίες, ε, θα πρέπει να τα ξανασυζητήσουμε και συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι στις συζητήσεις μας και στην προσέγγισή μας. Συζητώντας όμως την οδηγία θα πρέπει να παραμείνουμε και ρεαλιστές. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την προθυμία που εκδηλώσατε και εσείς συνάδελφοι και οι εκπρόσωποι της Επιτροπής και οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου. Και εμείς θέλουμε να έχουμε αρμονική συνεργασία. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ ωραία, σας ευχαριστώ για το χρονοδιάγραμμα. Ελέγχθησαν ήδη ορισμένα πράγματα. Κλείνω το σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης. Δεν ξέρω τώρα. Να αρχίσουμε το σημείο 11 ή να πάμε κατευθείαν στις ψηφοφορίες και να αφήσουμε μετά το 11. Ωραία. Σας παρακαλώ όμως, επειδή συνεχώς αναβάλουμε τη συζήτηση θεμάτων δεν θέλω, δεν ξέρω, θα αναγκαστώ να επανέλθω στις χθεσινές λύσεις όπου βάζαμε χρονογόρευσης. Τέλος πάντων, δεν μου αρέσει και αυτό. Ωραία λοιπόν. Α, ας προχωρήσουμε στις ψηφοφορίες. Έχετε τις κάρτες μαζί σας όλοι. Είναι έτοιμες οι κάρτες σας για τον αγώνα. Μπορούμε να αρχίσουμε. Πολύ ωραία λοιπόν. Αρχίζουμε λοιπόν βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης. Επί της διαδικασίας. Ματίας, παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να περιμένουμε νομίζω λίγο γιατί υπάρχουν συνάδελφοι που δεν έχουν φτάσει ακόμη. Για τις 10 προβλέπονταν οι ψηφοφορίες. Αρκετοί θα έρθουν μόνο για να ψηφίσουν. Κοιτάξτε την αίθουσα, είναι σχεδόν άδεια. Πέντε λεπτάκια. Εγώ λέω το ρολόι μου λέει 10. Δεν είναι 10. Ωραία. Ωραία, τότε λοιπόν αρχίζουμε το σημείο 11. Λοιπόν, δίνουμε το λόγο στη Ρίτα Κοχόλα για να αρχίσουμε το σημείο 11 της σημερινής διάθεξης, το οποίο θα διακόψουμε στις 10 και θα το συνεχίσουμε αργότερα. Παρακαλώ κυρία Κοχόλα. Για προσέξτε με. Ευχαριστώ. Αλλά καλό θα ήταν να έχω λίγο περισσότερο χρόνο από πέντε λεπτά. Ε, δεν μπορώ να τα πω όλα σε πέντε λεπτά. Καλά, θα επιταχύνω. Υποτίθεται ότι πρέπει να μιλήσω για την σύνοδο του Κανκούν, τη σύνοδο για τι κλιματικέ αλλαγέ στο Μεξικό. Ελπίζω να προλάβετε και να μπορέσετε να με ακούσετε. Ήμουν μέρο τη αντιπροσωπεία ε, που ήταν υπεύθυνη για το ψήφισμα που αφορούσε το Κανκούν με συγχωρείτε. Κυρίε και κύριοι, λίγη ησυχία. Δεν είναι δίκαιο. Δεν είναι σωστό αυτό. Είναι πολλοί αυτοί που πουσιάζουν, την τελευταία στιγμή, κάνουν πηγαδάκια. Κυρία Κορχόλα. The highly unsuccessful COP15 in Copenhagen μετά την τεράστια αποτυχία της Κοπενχάγης, το COP15 και τις προσπάθειες που έγιναν πέρσι. Πιστεύαμε ότι ο μηχανισμό για τι διαπραγματεύσει αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών είχε χάσει πλέον την αποτελεσματικότητά του και έφτανε στο τέλο τη ζωή του. Δεν έδινε αποτελέσματα. Ωστόσο, η Σύνοδο του Κανκούν στο τέλο μα εξέπληξε, διότι καταφέραμε να ολοκληρώσουμε και να περάσουμε τις, τα περισσότερα μέτρα που θέλαμε με, μόνο την, την Βολιβία να διαφωνεί. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό λοιπόν για τις διαπραγματεύσεις με περικλιματικών αλλαγών και υπάρχει ένα σημείο που παραμένει εκκρεμές. Βέβαια κάποιοι επικρίνουν τις διαπραγματεύσεις, όμως ο σύνοδος του Κανκούν έδειξε ότι σε επίπεδο ΟΗΕ 200 χώρε σε επιμέρου θέματα για τι κλιματικέ αλλαγέ, για το κλίμα, μπορούν να πετύχουν κάποια συμφωνία. Και ο Μεξικανό Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων, που προείδευσε σε κάποια συνάντηση, μπόρεσε να δημιουργήσει ε, ένα κλίμα εμπιστοσύνη, όπου είχαμε ανοιχτό διάλογο και αυτό ευχαρίστησε ιδιαίτερα κάποιε αναπτυσσόμενε χώρε όπω την Ινδία και την Κίνα. Οι βασικοί τομεί όπου πετύχαμε συμφωνία θα αναφέρω ορισμένους. Πρώτα απ' όλα αντιμετώπιση της αύξησης ε, της παγκόσμιας θερμοκρασίας κατά 2 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με την προβιομηχανική περίοδο. Έπειτα, οι συμφωνίες που θέλαμε να πετύχουμε και στην Κοπενχάγη για χρηματοδότηση ε, αναπτυσσόμενων χωρών από τους βιομηχανοποιημένες. Τρίτον, όλες οι χώρες δεσμεύτηκαν να καταμετρούν, να υποβάλουν εκθέσεις και να παληθεύουν τι εκπομπέ του. Αυτό ήταν μία από τι βασικέ προποθέσει για τι βιομηχανοποιημένε χώρε, ώστε και να χρηματοδοτούν ε, για αυτού του σκοπού τι αναπτυσσόμενε. Στη συμφωνία τη Κοπερχάγης συμφωνήθηκε τον Ιανουάριο του 2010 οι βιομηχανοποιημένε χώρε να να αναγγείλουν δεσμεύσει ε, για την αναχέτηση και τον περιορισμό των εκπομπών τους ώστε το 2020. Όλα αυτά ε, προσαρτήθηκαν στη συμφωνία που υπογράψαμε στο Κανκούν, όμω παραμένουν μη, μη δεσμευτικά τα μέτρα αυτά. Επίση, οι χώρε δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν τι διαπραγματεύσει του βάσει του πρωτοκόλλου του Κιώτο για τι μελλοντικέ του δράσει, ε, για τι βιομηχανοποιημένε χώρε. για το διάστημα 2008-2012 και μετά σε μια δεύτερη φάση για την περίοδο δεσμεύσεων από το 2013. Ε, όμως παραμένει σαφές ότι θα υπάρξει τελικά ένα κενό μεταξύ των δύο περιόδων. Η Ρωσία έχει πει ότι δεν μπορεί να αναλάβει μελλοντικέ ε, δεσμεύσεις και οι Ηνωμένε Πολιτείε ούτε στην πρώτη περίοδο δεσμεύσεων συμμετέχουν. Διότι δεν έχουν καν κυρώσει το πρωτόκολλο του Κιώτο. Και ο Καναδάς ανήγγειλε ότι το, το 2006 ότι αποσύρεται από το πρωτόκολλο του Κιώτο. Ενώ νωρίτερα είχε υπηκυρωθεί το πρωτόκολλο αυτό και είχαν συμφωνηθεί στόχοι περικόπη των εκπομπών. Έπειτα, οι αναπτυσσόμενες χώρες η αποψήλωση πρέπει να περιοριστεί στι αναπτυσσόμενες χώρες. Επίσης θα δημιουργηθεί μια ομάδα που θα εξετάζει τα θέματα αυτά. Ο μηχανισμός CDM για τις αναπτυσσόμενες χώρες ενισχύθηκε και θα περιλαμβάνει και τα προγράμματα CCS με πολύ αυστηρά κριτήρια όπως και τα προγράμματα CDM που είναι ήδη ένα πρώτο μικρό βήμα πρόοδου. Προκειμένου να προωθήσουμε την προσαρμογή ε, στους στόχους του Κανκούν, δημιουργήθηκε ένα σχετικό πλαίσιο και για να ανακεφαλαιώσω το κλίμα αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών σε σχέση με το, το σκηνικό μάλλον μετά το Κανκούν είναι ότι θα έχουμε πλέον ε, κάποιου στόχου περικοπή των εκπομπών, αλλά όχι δεσμευτικού για τι αναπτυσσόμενε ή για τι βιομηχανικοποιημένε χώρε. Θα μα λείψουν οι δεσμευτικοί στόχοι. Γιατί τελικά είναι έτσι τα πράγματα. Οι βασικότεροι ανταγωνιστές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ρωσία, η Ιαπωνία, οι Ηνωμένε Πολιτείε και ο Καναδάς είπαν όχι στην επόμενη περίοδο δεσμεύσεων του Κιώτο μετά το 2012. Εάν δούμε λοιπόν τις δεσμεύσεις αυτών των χωρών, βλέπουμε ότι η Ινδία, η Βραζιλία και η Κίνα, που είναι από αυτού που περισσότερο εκπέμπουν αεροθερμοκηπίου, δεν δεσμεύονται ούτε καν συμμετέχουν στην ομάδα αυτή. Και οι δράσεις του Προέδρου των ΗΠΑ και του Κογκρέσου θα ε, αρχίσουν μετά τις εκλογές. Ο κύριος Ομπάμα κάνει κάποια σταδιακά βήματα στην πολιτική για τις κλιματικές αλλαγές, αλλά τίποτα δεν έχει γίνει ακόμη στην πράξη. Εάν ε, οι διάδοχοι δεν κάνουν τίποτα περισσότερο, ή αν δεν αυξήσουν τι προσπάθειές του οι βιομηχανοποιημένε χώρε δεν θα επιτελεστεί πρόοδο. Οπότε τώρα θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα πιθανό σε επίπεδο ΟΗΕ οι χώρε αυτέ να κάνουν μονομερεί δηλώσει και να αναλάβουν μονομερό δεσμεύσει. Ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει το μοναχικό της δρόμο στις δεσμευτικές της, στα δεσμευτικά μέτρα και τις προσπάθειες περικοπής και μείωσης των εκπομπών. Το, 2000, το επόμενο κοπ θα γίνει τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο στην Νότια Αφρική, στο Ντέρμπαν, αλλά δεν αναμένουμε να ληφθούν εκεί σημαντικές αποφάσεις. Απλώς θα ανακεφαλαιωθούν και θα αποσαφινιστούν κάποια στοιχεία της συμφωνίας του Κανκούν. Σας ευχαριστώ πολύ που κάνατε την παρουσίασή σας τόσο ήρεμα και χαλαρά. Σταματούμε τώρα τη συζήτηση για το σημείο 11, την οποία θα συνεχίσουμε μετά τις ψηφοφορίες. Ε, Βλέπω ότι ήρθαν πολλοί συνάδελφοι εδώ για να ψηφίσουν στην αίθουσα, οπότε θα ήθελα να κάνω και κάποιες ανακοινώσεις. Ε, πρόσφατα, μάλλον και τούτη τη βδομάδα και στις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε πάρα πολύ φορτωμένες ημερήσεις διατάξεις. Πώς ε, ξεπερνούμε τα προβλήματα αυτά ή ορίζουμε χρόνο αγόρευσης, ένα-δυο λεπτά και ούτως ώστε να μιλήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι ή βγάζουμε θέματα από τη μυρίσια διάταξη. Τώρα η τρίτη δυνατότητα είναι να συγκαλέσουμε επιπλέον συνεδριάσεις. Θα πρέπει να σκεφτείτε αυτές, αυτά τα τρία σενάρια, να τα συζητήσετε στις πολιτικές σας ομάδες για να ε, πάρουμε μια κάποια απόφαση. Και αν, αν η λύση που προκρίνεται είναι να φορτώνουμε όλο και περισσότερο τις ημερήσεις διατάξεις μας, τότε κυρίες και κύριοι θα πρέπει και εσείς να δεχθείτε ε, να πειθαρχείστε σε συγκεκριμένους χρόνους αγόρευσης. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να ζητήσω πριν και μετά από τις ψηφοφορίες όπου μπαινοβγαίνει πολλοί κόσμος στην αίθουσα να κάνετε κάποια ησυχία διότι δεν είναι ούτε δίκαιο ούτε ευγενικό προς τους ε, συναδέλφους που μιλούν εκείνη την ώρα ε, να ε, γίνεται χάβρα να, να γίνεται θόρυβος μάλλον Λυπούμε, αλλά είμαι υποχρεωμένος να τα πω αυτά και καταλαβαίνω ότι δεν είναι δυσάρεστα αυτά που λέω. Αλλά αν θέλουμε να συνεχίσουμε να δουλεύσουμε καλά, αν δεν αυξήσουμε τον αριθμό των συνεδριάσεων και συνεχίζουμε να αυξάνουμε τα θέματα που βάζουμε στη μερίσια διάδεξη, άλλος, άλλη λύση δεν υπάρχει. Τώρα, αν έχετε άλλες ιδέες ή άλλες προτάσεις, ευχαρίστω να τις ακούσω. Ωστόσο, εδώ που βρισκόμαστε τώρα πρέπει να αυτοπιθαρχήσουμε να πειθαρχήσουμε όλοι και να αυτοπεριοριστούμε όλοι. Ζητώ συγγνώμη, αλλά θεώρησα ότι έπρεπε να λεχθούν αυτά για να είμαστε ξεκάθαροι ανάμεσά μας και για να έχετε κι εσείς κάπως μεγαλύτερη κατανόηση γιατί είμαι πολλές φορές τόσο αυστηρός. Λοιπόν, ψηφοφορίες. Πρώτη έκθεση του κυρίου Λάγκε, βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης. Υπάρχουν σωρό τροποποίησεις που καταθέτα, κατατέθηκαν, υπάρχουν και τρεις προφορικές. Λοιπόν, αρχίζουμε. Ε, λύση 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παρακαλώ τώρα. 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 56 υπέρ κατά συγγνώμη ξανά 56 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ ψηφίστε Εντάξει, πέρα τη ψηφοφορία. Ε, εγκρίνεται. Λοιπόν, 57 τώρα. Όχι, 58, συγγνώμη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Okay. 57, the uh, Το 57. Δεν νομίζω ότι ψηφίσαμε το 57, πρόεδρε. Also 57 im Kompromiss. Ναι, αλλά η 57 συμπεριλαμβάνεται στη συμβαστική λύση. Δεν χρειάζεται να την ψηφίσουμε. Λοιπόν, 65 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβασμός 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται επίσης συμβιβασμός 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 89 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 92 υπέρ Ποια την 89 αμφισβητείτε Ωραία ε, ηλεκτρονική επαλήθευση ψηφίστε την 89 Okay, okay. closed πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. 92 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ. 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 96 υπέρ κατά τσεκ 96 έλεγχος παρακαλώ πέρα στις ψηφοφορίες απορρίπτεται συμβασμός 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα 110 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβασμός 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβασμός 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 123 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 125 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 126 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 127 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 129 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 130 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 131 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 132 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 133 ως προσθήκη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 134 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 135 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 136 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 137 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 140 υπέρ κατά αποχές τσεκ 140 τσεκ 140 λοιπόν ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Μία επιπλέον βο... Ε, ψήφος για το ΕΛΚ. Όχι. Ναι. Much, ναι. Μία επιπλέον για το ΕΛΚ. Δεν ξέρω γιατί. Okay, okay, okay. okay, that's okay. And? Okay, that's it. No, it's okay, but we have no result. Okay. <laughs> yeah, adopted, thanks. Εγκρίνεται λοιπόν. 141 υπέρ. Ah, 142 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 143 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 144 υπέρ κατά κατά κατά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 Λοιπόν, συμβεσμόν 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 158 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 163 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 162 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 165 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 166 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβασμός 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 175 υπέρ ε, 170 ήταν αυτό, με συγχωρείτε, 171, 172 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 173 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 176 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 177 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 178 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 179 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 180 την 179 ωραία έλεγχος Ψηφίστε. Πέρας. Ένα, μία επιπλέον ψήφο ΕΛΚ. Ωραία, εγκρίνεται. 180 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 181 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 182 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβασμός 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 192 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Από το 153 λέει ο πρόεδρος 194 η 192 η 194 υπέρ κατά συγγνώμη 194 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 195 υπέρ κατά έλεγχος έλεγχος όχι την 194. Την 194. 195. 195. 195. 195. Okay? 195 ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα τη ψηφοφορία εγκρίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Συμβασμός 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 198 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβασμός 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 202 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 205 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 203 υπέρ κατά Uh, η 203 καταπίπτει, 204 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε τη 204 παρακαλώ. 204. Um, okay, closed. And adopted. Εγκρίνεται. Συμβασμός 14 υπέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 210 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβασμός 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 217 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 218 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβασμός 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 229 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ Λοιπόν, το πρώτο τμήμα καταπίπτει, δεύτερο τμήμα, 229, δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. We check. Really? You don't want? Miss Merkis. <laughs> Okay. 231. 231. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 18 με προφορική τροπολογία. Υπάρχουν ενστάσεις για την προφορική τροπολογία. From Alde. Miss Hall. Η κυρία Χολ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους συζητητές διότι μου επιτρέψανε αυτό να το περιλάβουμε και στο 18 είχαμε το θέμα της διατύπωσης, αλλά μόνο όταν είναι πλήρως συμβατό με τους στόχους της ανάπτυξης των οικονομικών συμφωνιών εταιρικής σχέσης. Υπάρχουν ενστάσεις για αυτή την ε, προφορική τροπολογία. Όχι. Λοιπόν, συμβασμός 18 υπέρ. <coughs> Κατά αποχές εγκρίνεται 244 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 247 υπέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 248 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 249 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 252 υπέρ Κατά. Λοιπόν, ξανά 252 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. 252. Ψηφίστε. And closed. Yeah, closed. And adopted. Εγκρίνεται. 253 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 254 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 255 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 257 Α, τη 255 Ωραία, ηλεκτρονική ψηφοφορία 255 Πέρας της ψηφοφορίας. ο, απορρίπτεται. Με σαφή πλειοψηφία κιόλα. 257 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 258 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 259. Τι αμφισβητείτε. Entschuldigung, war ein Bitte nimm es. ja klar, natürlich. 258 wird jetzt gecheckt. να το ελέγξουμε λοιπόν. 258, ψηφίστε. Ελπίζω να είχα δει και εγώ πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται στη Λοιπόν, 262 υπέρ κατά... Ε, 260, συγγνώμη. 261 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Zustimmung. 282 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 283 υπέρ κατά ξανά 283 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 284 υπέρ Ωραία, να ελέγξουμε τη 283 παρακαλώ. the board is and closed and Adopted. Εγκρίνεται. Τώρα 2.84 υπέρ. Κατά. 2.84 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.85 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.86 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.87 υπέρ κατά mm. έλεγχος τη 287 εγκρίνεται η 287 288 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 289 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 290 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβασμός 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 303 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 304 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 305 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 306 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 307 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 308 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 309 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 310 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 311 υπέρ κατά αποχές έλεγχος 311 εγκρίνεται 312 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3.14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3.15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3.17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 320 υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε. 320. Απορρίπτεται. 321 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 323 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ. Α, συγγνώμη. Number? Oral amendment from? Ms. oui. E Perhaps Ms. is oral amendment from you? Κυρία Τζαβέλα, υπάρχει. Ευχαριστώ, δεν θέλω, όχι, όχι, όχι. Ωραία, δεν χρειάζεται λοιπόν. Πάμε στην 3.25. Υπέρ. Χωρίς, χωρίς την προφορική τροπολογία κατά αποχές εγκρίνεται 326 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 327 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 328 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 λέει ο πρόεδρος. Α, συγγνώμη, 3.30 με προφορική τροπολογία. Ε. Ένσταση ουδές. 330 λοιπόν με την προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 331 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3.46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3.49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3.51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και 3.52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σεβασμό 22 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 3, 63 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 365 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 364 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 374. Α! Kompromiss 23. Συμβιβασμός 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ. 374. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 375. Έλεγχος 374. Ωραία. Ψηφίστε. Πέρας της ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 3,75 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 3,76 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται 3,77 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 3,77 Ωραία. 3,77 να ελέγξουμε. Πέρας της ψηφοφορίας. Ου, απορρίπτεται. 3,78. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3,79. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 24 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 383 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 384 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 387 με τροπολογία προφορική ένσταση για την προφορική τροπολογία έχει κανείς ουδής Πολύ ωραία λοιπόν. 3.87 με την προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 3.88 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 3.91 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 3.89 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 3.90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 392 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 393 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 94 υπέρ 90 ε, κατά αποχές εγκρίνεται 97 υπέρ κατά ε, εγκρίνεται 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβασμός 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 410 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβασμός 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 427 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 428 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ α καταπίπτει 434 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 34 434 in check vote is... Ωραία, έλεγχος 434. Απορρίπτεται. 4.36 περ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ωραία. Σοβαρά. Σοβαρά θέλετε επαλήθευση. Όχι. Ωραία. Συμβασμός 27 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 443 υπέρ. Κατά αποχές και αυτό τι εγκρίνεται 444 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 45 υπέρ κανείς ωραία κατά έλεγχος 4.45 Ψηφίστε. I must do it because 444 uh, was adopted. And there... Εγκρίθηκε η 444. Γι' αυτό πρέπει να ψηφίσουμε για την 445. Λοιπόν, ψηφίστε. Πέρας απορρίπτεται. Ωραία, τώρα 4.46 πέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4.47 υπέρ κατά αποχές 4.47 υπέρ κατά Excuse me, check 447 Ηλεκτρονική ψηφοφορία 447. Closed. And adopted. Εγκρίνεται 448 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 449 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 451 καταπίπτει ωραία 452 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβασμός 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 457 υπέρ κατά αποχές 467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 του 4, της 467 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 469 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 470 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 471 υπέρ κατά αποχές απορρι... Ε, εγκρίνεται mm -hmm. Συμβασμός 29 υπέρ κατά αποχές απορρι... Ε, εγκρίνεται 483 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 86 υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε την 486 ε, απορρίπτεται 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 88 υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε την 488 488 ψηφίστε πέρας ψηφοφορίας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 για το 5 αιτιολογική σκέψη α. Εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβασμός 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβασμός 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 με συγχωρείτε ήταν αυτό 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ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 2 έμπλ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 έμπλ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ήλτα 1 υπέρ 2 ε, κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ΙΜΚΟ 2 υπέρ κατά αποχές αρχίζουμε να αρχή 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ Α, έλεγχος. Ωραία, γιατί δύο. Γιατί δύο τη του Ψηφίστε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρία υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τέσσερα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πέντε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έξι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ α την 8 οκ 8 λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα καλύπτεται από το συμβασμό 6. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ κατά αποχές Είκοσι λοιπόν, ποιος είναι υπέρ, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ρέγγι 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ Τσεκ το 6. Ωραία. Ψηφίστε για την 6 της Ρέτζη. Εγκρίνεται. 10 υπέρ. Α, συγγνώμη. Το ξέχασα την 7. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά Συγγνώμη, να επαναλαμβάνουμε υπέρ της 15 κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα επιτέλους η τελική ψηφοφορία Do your very best also ähnlich and closed closed and adopted εγκρίνεται λοιπόν συγχαρητήρια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 Adopted. Εγκρίθηκε. Πούντς. Μπράβο, συγχαρητήρια κύριε Κλάντε. Τέτοιου είδους voting list θέλουμε στο μέλλον, ε. Mm. Όχι σαν του Λάγκε. Λοιπόν, προχωρούμε. Στη... Συμβιβασμός 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τέσσερα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Έξι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Εφτά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Εννιά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβασμός 2 υπέρ κατά αποχές Συμβασμό 3 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχέ ε, εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται 24 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά για να το ελέγξουμε δεύτερο τμήμα υπέρ. Εγκρίνεται. 25. Ως πέρα, υπέρ. Κατά. Ένα λεπτό. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ωραία. Έλεγχος. Παρακαλώ. Πέρα στις πληροφορίες. Εγκρίνεται. 26 πέρ. Κατά. Αποχές. Ξανά, ε, 26 πέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 27 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 σε τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα καταπίπτει. 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ κατά αποχές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 αποχές έλεγχος έλεγχος ηλεκτρονικός έλεγχος εγκρίνεται τελική ψηφοφορία α συγγνώμη την 54 ξέχασα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Final vote υπέρ. Ε, ψηφίστε με συγχωρείτε. Can begin? Yeah. Yeah. Vote is open. And the vote is closed and is adopted. Thank you. Thank you, Rapporteur. Εγκρίνεται. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον εισηγητή. Προχωρούμε Ξαναγυρνάμε στο σημείο 1. Κλείσα, τελειώσαμε τις ψηφοφορίες. Ξαναγυρνάμε στο σημείο 11 τη ημερησία διάταξη. Ησυχία κατά την έξοδο όμω. Η κυρία Καβάλιο ζητεί το λόγο. Για το 11 φαντάζομαι. Η κυρία Καβάλιο, έχετε το λόγο. Oh, Should I start? let us a chance to start. Παρακαλούμε αφήστε μας την ε, δυνατότητα να συζητήσουμε. Η μόνη που θέλω να ακούγεται στην αίθουσα τώρα είναι η κυρία Καρβάλιου. Uh, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ είχα συμμετάσχει στην αντιπροσωπεία που πήγαμε στην Κακούν στο COP16 και είχα συμπροεδρεύσει σε εκείνη την ομάδα για τα βιομηχανικά θέματα και από το 98 και μετά πάω πάντοτε στα COP16 οπότε και θεώρησα ότι η Κακούν είναι μία από τις πιο αποδοτικές συναντήσεις ε, λόγω της καλής Μεσικανικής Προεδρίας, ο Πρόεδρος Επιμελητίας, περιεχομένο, ε, διεύθυνση των εργασιών, διαφάνειας, αποτελεσματικότητα, σε αντίθεση με τις προηγούμενες κόπ. Ας πούμε την κόπ 16 την προηγούμενη, στην Pyongyang. Τώρα Έχουμε το θέμα δύο εγκρίσεων αποφάσεων της ΚΟΠ που αντίθετα με ήταν στο παρελθόν τώρα έχουμε μια μακρόπνοη απόφαση η μία φορά τη σύμβαση και η άλλη φορά το πρωτόκολλο του Κιώτο. Να συνεχίσω. Λοιπόν, σα επισημαίνω συνάδελφοι ότι δεν είχα συμμετασχεί και τόσο πολύ σε αυτές τις ε, διαπραγματεύσει, έχουμε δύο παράλληλε. Πρώτα-πρώτα, μία σύμφωνα με την σύμβαση και την ένταση με το πρωτοκόλλο του Κιώτο, οπότε και βέβαια η Αμερική λαμβάνει, μόρα, λαμβάνει μέρος ε, στη μία και όχι στην άλλη, και όχι στο Κιώτο δηλαδή. Και όταν είπαμε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα στις διαπραγματεύσεις για τη Ρωσία η οποία δεν έχει προσχωρήσει στη δεύτερη περίοδο του πρωτοκόλλου του Κιώτο, αυτό έγινε κατά τι διαπραγματεύσει του Κιώτο και όχι τη μακρόπρόθεσμε. Οπότε, στο COP16 είχαμε πάρα πολύ δυνατό πρόοδο. Ιδίω όσον αφορά τι ε, διαπραγματεύσει για την ε, σύμβαση. Και έχουμε λοιπόν, επομένω ε, ε, αυτή την παράλληλη διαδικασία, η οποία ήταν αρκετά συλλογημένη, διότι πριν το COP16 το Κιώτο προχωρούσε πιο δύσκολα από ό,τι η σύμβαση. Οπότε ήταν πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των δύο και να είναι δυνατόν να προχωρήσουμε όσον αφορά τις ε, διαπραγματεύσεις για την σύμβαση, γιατί εκεί παρίσταντο όλοι περίπου 194. Και είχαμε μόνο μια υπομάδα για το Κιώτο. Η υπομάδα χωρών. Οπότε, ολοκληρώθηκε η ΚΟΠ με δύο αποφάσεις, οι οποίες ενεκρίθησαν. Μόνο η Βολιβία κατεψήφισε. Όλοι οι άλλοι ενέκριναν, επιψήφισαν και χειροκρότησαν η χειρά την Προεδρία. Και από ό,τι ξέρω αυτό γίνεται για πρώτη φορά. Η Σάδος σας ανέφερε τα βασικότερα και επομένως από τα βασικά είναι ότι έτσι υπήρξε η δέσμευση. στη συνέχιση των όσων στην Pyongyang και στο ΝΟΙΕ. Κάναμε όμω ζητήματα πρόοδο όσον αφορά το ταμείο κλίμα, το πακέτο για τα δάση, την τεχνολογική προσαρμογή κλπ. Οπότε, εν κατακλείδη και πάλι θεωρούμε ότι θα πάνε καλά τα πράγματα στο, στο, και υπάρχει κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πιο θετική τώρα η στάση και της Αμερικής και της Κίνας. Επίσης, να αναφέρω την Ευρωπαϊκή Προεδρία, η οποία ήταν πάρα πολύ αποτελεσματική και από πλευράς Κομισιόν και πλευράς Βελγικής Προεδρίας. Επίσης και οι επαφές μας τα πήγαν πάρα πολύ καλά, ο Σκηνοβούλη και γίνανε συγκεκριμένα βήματα σε πάρα πολύ σημαντικούς τομείς, οπότε θα έχουμε έτσι μια γενική συμφωνία θα υπάρχει στέρη βάση, αφετηρία για διαπραγματεύσεις για να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε ε, στην επόμενη κόπ στην Νότιο Αφρικανική Δημοκρατία. Στις 12 παρατέταρτο θα έρθει ο υπουργό. Και έχουμε άλλα θέματα τώρα πριν από αυτό στην Μεσδιαδίξη, οπότε παρακαλώ συνάδελφοι. Ένα λεφτάκι μόνο. Uh, thanks, uh, chairman. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα ξεπεράσω τα δύο λεπτά, απλώ σε όσα είπαν οι συνάδελφοι για τα αποτελέσματα της ΚΟΠ, να πω ότι καλό είναι να έχουν μια ιδέα και συνάδελφοι που δεν ε, ήταν εκεί. Τι είδους πρόγραμμα εξετάσαμε. Τι συζητήθηκε εκεί. Συγκεκριμένα, Πήγαμε ως εκεί με 12 μέλη της Επιτροπής Ήτρε και όπω είπε η κυρία Καρβάλιο συμμετείχαμε σε τρεις ομάδες εργασίας για την ε, μεταφορά τεχνολογιών και τη βιομηχανία η πρώτη, για την αποψήλωση η δεύτερη και για τους μηχανισμούς αγοράς και διεθνεί οργανισμού η τρίτη. Ήταν πολύ θετική η εμπειρία μας ως προς την ανταλλαγή απόψεων και είχαμε αρκετές διμερείς συναντήσεις. Όχι μόνο με τους Αμερικανούς, αλλά και τους Ιάπωνες και τους Μεξικανούς και με Βραζιλιάνους. Ήταν πολύ ενδιαφέρον όχι μόνο η ανταλλαγή απόψεων, αλλά και η ευκαιρία που μας δόθηκε να προωθήσουμε τις δικές μας απόψεις, να εξάγουμε των εισαγωγικών το ευρωπαϊκό μοντέλο και την ευρωπαϊκή προσέγγιση. Αυτά κάναμε και με την αμυντική μας πολιτική για να την πω έτσι. Δηλαδή είχαμε από τη μια της ομάδας εργασίας και παραλλήλως δύο εργαστήρια τα οποία ήταν ανοιχτά σε όλους τους συμμετέχοντες στην ε, Σύνοδο ΚΟΠ. Εκεί λοιπόν υπήρχε ιδιαίτερη συμμετοχή. Ένα από αυτά τα εργαστήρια ασχολείται με την μεταφορά τεχνολογιών και την ενεργειακή αποδοτικότητα όπου προείδρευε ο κύριος Λάινεν ε, της Επιτροπής ΕΝΒΗ και έπειτα ένα άλλο εργαστήριο για την εκπομπή αερίων από την αυσιπλοεία και την αεροπλοεία. Εκεί επίσης είχαμε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Το αποτέλεσμα λοιπόν της COP16, όπως είπε η κυρία Καρβάλιο και η κυρία Κορχόλα, ήταν ε, ενδιαφέρον. Δεν θα τα επαναλάβω, απλώς για να ολοκληρώσω πρόεδρε, να πω ότι ευχαριστώ ιδιαίτερα στο προσωπικό της Επιτροπής ΕΝΒΗ και της Επιτροπής Ήτρε και το Γιώργιο και τους υπόλοιπους συναδέλφους της Γραμματείας που ήταν πάντοτε στη διάθεσή μας με την τεχνογνωσία τους. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερος, κυρία Ματίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και εγώ να προσθέσω τις δικές μου ευχαριστίες και προς τους εκπροσώπους της ε, Επιτροπής, προς τους υπαλλήλους μάλλον της Επιτροπής μας που έκαναν εξαιρετικό έργο. Όπως είπε και η κυρία Κορχόλα, ε, που σωστά αξιολόγησε τη σύνοδο του Κανκούν. Θα προσπαθήσω και εγώ να παραμείνω στο ένα λεπτό όπως μας ζητήσατε και να πω ότι είναι μακρύς ο δρόμος μας μέχρι την Νότια Αφρική. Ιδίως σε δύο τομείς, μεταφορά τεχνολογιών και τα ζητήματα της ενέργειας. Εκεί πολλά πρέπει να πούμε και θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ενεργά σε αυτήν την Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο για να προσπαθήσουμε στην Νότια Αφρική να έχουμε δεσμευτικούς πλέον στόχους. Και βεβαίως να αναλάβουν τις ευθύνες τους όλες οι χώρες που υπέγραψαν τη συμφωνία. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, 15 Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών. Να δώσω το λόγο στον κύριο Τσίτσεστερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή, οι δύο δηλαδή εκθέσεις, αφορούν τον οργανισμό για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών. Όπως θα θυμούνται κάποιοι συνάδελφοι, Είχαμε ασχοληθεί με την ύπαρξη μιας τέτοιας επιτροπής στην προηγούμενη θητεία. Αφού συζητήσαμε, προβλέψαμε παράταση της θητείας της Επιτροπής εκείνης. Τώρα μας έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύο προτάσεις. Η μία είναι επί της ουσίας αναθεώρηση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του οργανισμού. Η άλλη μια πρόταση για την ε, πλαισιωμένη παράταση της θητείας της Επιτροπής αυτής διότι θα λήξει η εντολή της Επιτροπής αυτής τον Μάρτιο του 2012 προτείνεται λοιπόν να παραταθεί η λειτουργία της ως το Σεπτέμβριο του 2013 όπως έχει πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό είναι ένα μέτρο πρόληψης εφόσον δεν προχωρήσουμε τελικά τόσο γρήγορα όσο θα ήθελαν, ε, στην επί της πρόταση που αναθεωρεί τον κανονισμό. Οπότε, Πρόεδρε, ήθελα να ευχαριστήσω τους χιώδης εισηγητές. Είχαμε ήδη δύο συναντήσεις. Στην πιο πρόσφατη είχαμε μια χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων για τα ζητήματα που μας απασχολούν εδώ να πω ευθύς εξ αρχής ότι υπάρχει εδώ ένα βασικό ζήτημα που δεν καλύπτεται από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που όμως θα πρέπει να το επιλύσουμε, διότι μας απασχόλησε και μας ενόχλησε προηγουμένως όταν εξετάζαμε τον κανονισμό αυτού του οργανισμού πάλι. Και αυτό είναι η έδρα, το που θα τοποθετηθεί αυτός ο οργανισμός ειλικρινώ αυτό είναι καθοριστική σημασία. Προκειμένου να ε, λειτουργήσει αποτελεσματικά αυτό ο οργανισμός και ω προ τα κονδύλια που θα απορροφήσει. Πρέπει να εκφράσω εδώ την ε, δυσαρέσκειά μου που θα πρέπει να επιμείνω σε αυτό, αλλά μετά από αριθμό μελετών, ιδίω στη Βουλή των Λόρδων, στο κράτο μέλο από το οποίο προέρχομαι, επικεντρωθήκαμε Ακριβώς το θέμα της έδρας αυτού του οργανισμού. Βρίσκεται στην Κρήτη. Υπέροχο το νησί. Το επιβεβαιώνω. Έχω πάει εγώ εκεί. Διακοπές. Όμως είναι και πολύ μακριά. Είναι μεγάλο το ταξίδι για να πάει κανείς. Αυτός είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει την αποτελεσματική λειτουργία του οργανισμού και βεβαίως τις συνθήκες διαβίωσης του προσωπικού. Ένα άλλο θέμα εδώ είναι ότι αυτό πρέπει να επιληθεί διότι οι λεπτομέρειες, ε, μάλλον οι υποχρεώσεις που προβλέπονταν από τη συμφωνία του κράτους υποδοχής δεν ε, πληρώθηκαν πλήρως. Και αυτό είναι ένα θέμα. Οι ελληνικές αρχές αντιμετωπίζουν δυσκολίες αυτή την περίοδο. Οι δεσμεύσει λοιπόν που είχαν αναλάβει δεν έχουν πληρωθεί. Ε, Με την πρόταση λοιπόν αυτή έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε τα θέματα που μας απασχολούν. Πρόεδρε, εδώ έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων ε, σε, πρώτε, σε πρώιμα στάδια έτσι κι αλλιώς. Δεν θα περάσω σε περισσότερες λεπτομέρειες, απλώς θέλω να πω ότι προτείνω να καταβάλουμε προσπάθειες ώστε η πρώτη μας πρόταση για παράταση της θητείας, για αυτή τη σύντομη παράταση της θητείας, της εντολής της Επιτροπής, να δοθεί μέσω της ταχείας διαδικασίας. Να είμαστε όσο το δυνατόν ε, πιο ταχείς, ώστε να στείλουμε έτσι και ένα σαφές μήνυμα στο προσωπικό του οργανισμού, ότι του στηρίζουμε. Θέλουμε να συνεχίσουν το έργο τους. Απλώς θέλουμε να υπάρξει κάποια αναδιάρθρωση και θέλουμε χρόνο να δούμε πώς ακριβώς θα γίνουν τα πράγματα. Οι αρμοδιότητές τους, ο ρόλος τους είναι προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Είναι θέματα στα οποία πρέπει να βρούμε λύσεις. Ο οργανισμός αυτός ασχολείται με ζητήματα που τα θεωρούμε άκρο σημαντικά. Ιδίω οι οργανισμοί των κάτω μελών που ασχολούνται με το διαδίκτυο, την ασφάλεια των πληροφοριών και των δικτύων, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Αυτό είναι ο όρο. Cyber security. Εάν θέλουμε λοιπόν να αλλάξει ο ρόλος του οργανισμού, θα πρέπει να φροντίσουμε να μην επικαλύπτει ωστόσο το τι κάνουν και εθνικοί οργανισμοί. Θέλουμε να έχει ευρωπαϊκή αξία και νόημα ο οργανισμός στη λειτουργία του. Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της θίγει αρκετά ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του οργανισμού Κανένα από αυτά όμως δεν αφορά την έδρα. Γι' αυτό εγώ την είπα πρώτη-πρώτη. Αναφέρουν την ε, διαφορά και τον κατακαιρματισμό των εθνικών προσεγγίσεων, την ε, ευρωπαϊκή διαδικασία έγκαιρης αντίδραση τις περιορισμένες γνώσεις για τα προβλήματα διασύνδεσης, την έλλειψη ενημέρωσης και την ασφάλεια των πληροφοριών, τους σχετικούς κινδύνους, τις απειλές, ε, την διεθνή διάσταση της ε, ασφάλειας στο διαδίκτυο και των σχετικών προβλημάτων, τις ανάγκες για τα πρότυπα συνεργασίας προκειμένου να διασφαλίσουμε κατάλληλη πολιτική υλοποίηση και την ανάγκη για αποτελεσματικότερη δράση κατά των εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο. Αυτή είναι η άποψη της ασφάλειας από την, άποψη από την πλευρά των πολιτών. Και αυτά τα προβλήματα εντοπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά ε, αναλύονται περισσότερο στην επί της πρότασή της. Δεν θα επιλύσουμε όλα αυτά τα ζητήματα σήμερα το πρωί βεβαίω. Όμως, Θα ήθελα να ζητήσω από τους συντονιστές να προβλέψουμε μια μήνυ ακρόαση για το θέμα αυτό. Να έρθουν εξωτερικοί εμπειρογνώμονες για να μας ε, παρουσιάσουν στοιχεία και απόψεις ανεξαρτήτως των στοιχείων που μας ε, παρέχει η Κομισιόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, έχει κάνει τεράστιο έργο, αλλά βρίσκω ότι χρήσιμο θα τα να έχουμε για μια μήνυα ακρόαση. Και επειδή έχουμε αυτές τις δυνατότητες, να ζητήσουμε από την Επιτροπή μια σύντομη μελέτη για το θέμα αυτό, έτσι άμεσα, ώστε να έχουμε και μια άλλη προοπτική για το θέμα. Εγώ είχα μια προκαταρκτική συνάντηση με τους εκπροσώπους της Ουγγρικής Προεδρίας και εκεί εκφράστηκε η ελπίδα ότι θα ελοκληρώσουμε την εξέταση του θέματος αυτού επί της Προεδρίας τους. Μπορεί δυστυχώς να τους απογοητεύσω βέβαια, διότι το θέμα αυτό είναι σοβαρό. Είναι σοβαρό το Πρέπει να το δούμε με μεγάλη προσοχή. Και αν θέλουμε να το δούμε σε όλες τις λεπτομέρειες με προσοχή, δεν μπορούμε να δεσμευτούμε τώρα ότι θα ολοκληρώσουμε την πρόταση αυτή και την εξετασή της πριν το δεύτερο εξάμεινο της χρονιάς. Πρόεδρε, αυτά ούτως ή θα τα ξανασυζητήσουμε και στους συντονιστές. Και δεν θέλω να επιμείνω σε αυτό τώρα. Για την ώρα νομίζω ότι είπα αρκετά, ίσως κάποια να τα παρέλειψα, όμως ε, είμαι βέβαιος ότι οι συνάδελφοι θα τα θίξουν και θα τα σχολιάσουμε. Θα παραχωρήσω λοιπόν το λόγο στους υπολείπους για να ακούσω τι έχουν να πούν και οι συνάδελφοι. ich bitte nochmal, dass wir uns ein bisschen kurz fassen. Christian Ehlert, Frau Tikau. Παρακαλώ, να είστε σύντομοι, λέει ο Πρόεδρος. Ο επόμενος όποιος είναι. Ποιος είναι. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και τον Ούγγρο Υπουργό. Κρίστιαν. Πρόεδρε, πρώτα-πρώτα, για να δούμε την γενικότερη κατάσταση. Νομίζω ότι ε, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, ουσιαστικά συμφωνούμε. Είναι σημαντικό αυτό. Επίσης, θα πρέπει να ξέρουν, Συμβουλή Κομισιόν, ότι εμείς εδώ είμαστε αποφασισμένοι και θέλουμε να υπάρξει υπηρεσία λειτουργική, αποδοτική. Δεν είναι θέμα οργανωτικό, είναι πολιτικό. Έχουμε όλα αυτά τα θέματα τα οποία ε, στην πράξη ανακύπτουν. α πούμε είχαμε αυτή την επίθεση που έγινε την περσμένη εβδομάδα. Ε, επομένως λοιπόν, είναι θέμα του να προστατευτεί η πολιτική περιβάλλοντος που υφίσταται επιθέσεις επομένως. Αυτό θέλουμε. Θέλουμε αυτό να ρυθμιστεί που είναι θέμα και πολιτικό. Να δούμε επομένω το θέμα της έδρας. Υπάρχει εδώ συμφέρον και ενδιαφέρον πλευράς της χώρας. Ένα αυτό. Άλλο τώρα. Έριξτε μια ματιά. Βρισκόμαστε τώρα στο 0 όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και στο 10 είναι άριστα 100%. Οπότε και έχετε τα σχετικά εκτελεστικά δικαιώματα και η Κομισιόν τώρα λέει να πάμε στο επίπεδο αποτελεσματικότητας 4. Άρα προς τα εκεί θα πρέπει να κινηθούμε. Πάρα πολύ θετικά όλα αυτά. Φυσικά επιδέχεται βελτίωση η πρόταση. Η κυρία Γκρός ανέλαβε την ευθύνη για αυτό το σημαντικό θέμα. Πάντως εδώ έχουμε τρία τα οποία λείπουν από την έκθεση. Πρώτα-πρώτα από πλευράς οργανωτικής Μιλούμε για κάθετη οργάνωση. Όμως, για την ίσα και το GRC Υπάρχουν, υπάρχει εκτό από την ε, ε, ΕΝΙΣΑ και το GRC. Η ΕΝΙΣΑ έχει οριζόντιες σχέσεις με κάποιους άλλους οργανισμούς, αλλά με την Κομισιόν έχει κάθετες σχέσεις. Λοιπόν, ε, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο περι, δεν περιγράφονται τόσο απλά όπως λέγεται εδώ και μια και ε, πληρώνουμε ένα τόνο λεφτά για, τις, ε, για την ασφάλεια στο διαδίκτυο θα πρέπει να είμαστε σαφείς. Εδώ δηλαδή η, η έκθεση σχετίζεται, αναφέρεται στη σχέση του οργανισμού με, με την Κομισιόν αλλά υπάρχουν όμως οι σχέσεις, και οι σχέσεις του οργανισμού με άλλα προγράμματα και άλλους οργανισμούς και αυτές δεν περιγράφονται. Κάτι τι άλλο. Ποια είναι οι σχέσεις με τους άλλους ε, διεθνείς οργανισμούς. Το Κογκρέσο το Αμερικάνικο έχει κάποιο δικό του οργανισμό που φτιάχτηκε πριν από ένα χρόνο. Ε, ξεκίνησαν ε, συζητήσεις για το σύνολο των κανονιστικών διατάξεων του cyber security και αυτό αυτός ο οργανισμός είναι ο διαπραγματευτής. Πώς συνδέεται ο οργανισμός με τον Αμερικάνικο οργανισμό. Και ένα τρίτο θέμα που λείπει είναι το θέμα των, της κρίσιμης υποδομής στην Ευρώπη. Έχουμε, οι Υπουργοί Εργασίας πήραν μια απόφαση ε, στην οποία λένε ότι θα καθίσουν να σκεφτούν κατά πόσον η, το IT είναι κρίσιμη υποδομή. Για μένα είναι εκπληκτική η απόφαση αυτή η ασφάλεια στο τομέα της πληροφορικής στο κυβερνοχώρο είναι πολύ σημαντική και η ΕΝΙΣΑ και οι σχετικοί οργανισμοί που ασχολούνται με την ασφάλεια είναι η μία πτυχή του θέματος. Υπάρχουν και οικονομικά θέματα που σχετίζονται με αυτή την υπόθεση και το θέμα δεν είναι τόσο αν για την ασφάλεια θα την εξασφαλίζουν ε, κρατικά κονδύλια ή κάτι τέτοιο. Το θέμα είναι τι γίνεται από οικονομικές απόψεις και που, είναι, που βάζουμε κάποιες κόκκινες, κάποιες διαχωριστικές γραμμές για το τι μπορούν να κάνουν ιδιωτικές επιχειρήσεις. Πώς ρυθμίζεται και πώς εξασφαλίζονται ορισμένα πρα... η τήρηση ορισμένων αρχών στον ιδιωτικό τομέα της ε, πληροφορικής. Νομίζω ε, ότι αυτά τα τρία πράγματα λοιπόν λείπουν ε, από την έκθεση εμείς νομίζουμε ότι θα έπρεπε να περιλαμβάνονται και είμαστε ε, διαθέσιμοι να συζητήσουμε τα θέματα αυτά με την Κομισιόν. Τώρα <coughs> θα θέλαμε επίσης να πιστεύουμε ότι μπορούμε να έχουμε να καταλήξουμε σε μια ε, σαφή ισχυρή θέση από πλευρά κοινοβουλίου αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δώσουμε κάποιο χρόνο και στον εισηγητή. Εμεί θεωρούμε ότι είναι υψηλή πολιτικής σημασίας το θέμα αυτό και ιδιαίτερα το θέμα των υποδομών όπως είπα προηγούμενα, γιατί πιστεύουμε ότι η Ευρώπη στο σύνολό της δεν έχει αποτελεσματικές ε, υποδομές. Τι κάω. Uh, Ευχαριστώ πρόεδρε, να ευχαριστήσω τον κύριο Τσίτσεστερ γιατί συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά. Όπως είπαν και οι προηγούμενοι, πάρα πολύ σημαντικό το κοινοβούλιο να είναι ισχυρό στις διαπραγματεύσεις. Αυτές οι διαπραγματεύσεις θα κάνουμε με Συμβούλιο και Κομισιόν. Για να δούμε τι μορφή θα λάβει τελικά αυτή η υπηρεσία. Και συζητάμε τώρα για επέκταση, αλλά τέλος πάντων το θέμα είναι τι θα γίνει με κάποιο μακρόπνοη ασφάλεια. Να δούμε επίση πώ θα διαπραγματευτούμε με του διεθνεί μα εταίρου για τα θέματα τη ε, ασφάλεια και τα δίκτυα. Οπότε το πιο σημαντικό είναι να παραταθεί η ισχύς του κανονισμού για να μπορέσουμε να καλύψουμε ό,τι θέλουμε και εγκαίρως γιατί αρχά του 2012 θα λήξει αυτή η εντολή και αν δεν κάνουμε τώρα την παράταση θα υπάρξει χρόνος να γίνει η συζήτηση στα σοβαρά των αρμοδιοτήτων της νέας υπηρεσίας. Άρα θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με αυτή την πενταετή παράταση, όμως από την άλλη θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση όσον αφορά ευθύνες, αρμοδιότητες Πάρα πολύ σημαντικό αυτό και θα πρέπει να γίνει με σωστή συζήτηση. Τώρα όσον αφορά τους εμπειρογνώμονες την πλαισίωση της Νίσα θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει μετά την πενταετία. Αυτά για την Νίσα. Θα πρέπει να δούμε πώς θα αποκτήσει αξιοπιστή αυτή η υπηρεσία. Και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε πώς θα συντονιστούν και οι, του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα. Άρα πάμε μετά την πενταετία. Γι' αυτό σας λέω ότι μπορούμε όλα αυτά να τα δεχτούμε. Να πάμε μετά την πενταετία και να σκεφτούμε τελικά ποια θα είναι η τελική μορφή αυτής της υπηρεσίας και ποιε θα είναι οι τελικές αρμοδιότητες. Αν θα υπάρχει υπηρεσία που θα φροντίζει την κυβερνοασφάλεια, και θα κάνουμε σε προοπτική 15 20 ετή για να είναι μια υπηρεσία ισχυρή και αξιόπιστη και να έχει αρκετές αρμοδιότητες. Thank you. Uh, thank you. As, um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και όλους για την έκθεση αυτή. Να εκφράσω τη στήριξή μου για την προσέγγιση του κυρίου Τσίτσεστερ Συμφωνώ ότι χρειαζόμαστε μια προσέγγιση ταχύς διαδικασίας και ότι μπορούμε να προβλέψουμε την υπεραραία τάση της θητείας ως το 2013. Εδώ καλωσορίζω το γεγονός ότι η Επιτροπή μας θα πρέπει να έχει το χρόνο για να εξετάσει τις λεπτομέρειες της λειτουργίας του οργανισμού αυτού και πώς θα, πώς θα αναμορφωθεί εντολή για τις αρμοδιότητες του οργανισμού αυτού. Δεν θέλω να πω τώρα τι λεπτομέρειε τη όλη συζήτηση. Απλώ να κάνω μια-δυο παρατηρήσει για τη μελλοντική λειτουργία του οργανισμού. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να καθορίσουμε πώς οι πληροφορίες για τις εταιρικές σχέσεις δημόσιο-ιδιωτικού τομέα ε, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού θα ανταλλάσσονται. Ποιο θα είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών, εάν θα είναι πιο ακριβής οι κατάλογοι που θα προβλέψουμε και να έχουμε και την μέγιστη δυνατή ασφάλεια για τις επενδύσεις. Επίση, φαίνεται ότι η ασφάλεια γίνεται μια από τι πρώτε προτεραιότητε και για τι κρατικέ προμήθειε και για τα συστήματα ανταλλαγή πληροφοριών και τα δίκτυα τα κυβερνητικά. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχυθεί η ασφάλεια με μια κοινή δομή. Να υπάρχουν ανακοινώσει και ενημέρωση για όλα τα σημαντικά γεγονότα. και να ορίσουμε μια σχέση συνεργασίας διεθνή με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ίσως τα κάτι μέλη να μην ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την ανταλλαγή τέτοιων ευαίσθητων πληροφοριών, όμως τέτοιες πτυχές οφείλουμε να τις εξετάσουμε για να δούμε κατά πόσο είναι εφικτά όλα αυτά και να υπάρξει ικανοποιητικό συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών. Ναι. Πιστεύω ότι υπάρχει σαφής ανάγκη για τη λειτουργία της ΕΝΗΣΑ και θα πρέπει η λειτουργία του οργανισμού αυτού να, να γίνει λιγότερο γραφειοκρατική, περισσότερο αποτελεσματική. Και ίσω να συμμετάσχει εδώ και ιδιωτικό τομέα. Θα δούμε τη μελέτη που ζήτησε ο κύριο Τσίτσεστερ από του ε, υπευθύνου. Και τέλο, αυτό που θέλω να πω για το θέμα της έδρας της ΕΝΗΣΑ. Εφόσον γίνει η συζήτηση για την έδρα, πρέπει να σκεφτούμε το εξής σε τι συγκεκριμένα γεγονότα μπορούμε να βασιστούμε, στοιχεία μάλλον, ε, τι πληροφορίες μπορούμε να συλλέξουμε και πώς δεν θα χάσουμε από τις προτεραιότητές μας τη βασική προτεραιότητα, το βασικό στόχο, να παραμείνει καλή και να βελτιωθεί η λειτουργία της ΕΝΗΣΑ. Giles, θέλεις πάλι το λόγο? Δεν ξέρω αν θέλει να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτή τη φάση, Πρόεδρε. Θα την παρακαλούσα να μην παρέμβει, διότι χρόνο δεν έχουμε. Αλλά τέλος πάντων. Ένα λεπτό, ένα λεπτό για την Κομισιόν, λοιπόν. Λυπάμαι, γιατί έχουμε και προσκεκλημένους, ε, οι οποίοι έρχονται και περιμένουν. Λοιπόν, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τα μέλη του Κοινοβουλίου που έλαβαν το λόγο. Βεβαίω, αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην ενίσα. και Βεβαίω πρέπει να προβλέψουμε δίχτυα ασφαλεία για την λειτουργία με την παράταση τη ε, θητεία. Όπω ξέρουμε, εκπνέει η θητεία αυτή το Μάρτιο τη επόμενη χρονιά. Συμφωνούμε με τις προτάσεις σας ως ηγετού και εμείς θα συνεισφέρουμε στις συζητήσεις σας όπως θεωρείτε ότι σας χρειάζεται. Σα Σας ευχαριστούμε, Τζαίλ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις επικοδομητικές τους παρατηρήσεις και την Επιτροπή για την επικοδομητική της παρέμβαση. Οι συνάδελφοι και σε επίπεδο συντονιστών ελπίζω να συμφωνήσουμε με την πρόταση για μήνυα ακρόαση και για τη μελέτη που ζητήσαμε. Και θα επανέλθουμε ξανά με στη χρονιά. Ευχαριστούμε. Προθεσμή για την υποβολή τροπολογιών 28 Ιανουαρίου στις 10 το πρωί. Μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε. Μόνο για την παράταση της ε, λειτουργίας μιλάμε, έτσι. Λοιπόν, σημείο 16 στην ημερήσια διάταξη. Έχουμε τον κύριο Κάρλο Ντεσδορίδες, εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής για το σύστημα GNSS. Ε, με μεγάλη χαρά σας έχουμε σήμερα εδώ. Θα σας δώσω την ευκαιρία να συστηθείτε και ίσως να ακούσετε και κάποιες ερωτήσεις για να απαντήσετε. Συγχωρήστε μας, δεν ήμασταν και τρευγενικοί μαζί σας σήμερα το πρωί. Ήταν πολύ φορτωμένη η μερίσια διατάξη μας, δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Έχετε λοιπόν κατευθείαν το λόγο. So, Mr. Chairman, uh, Πρόεδρε, μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου σε αυτή μου την πρώτη επίσκεψη στην Επιτροπή σας Ήτρε να ξεκινήσω λέγοντας ότι γνωρίζω πολύ καλά το νέο θεσμικό αρχιτεκτόνημα που ε, εγκαθιδρύεται με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ξέρω τον ε, σημαντικότατο ρόλο που διαδραματίζει πλέον το Κοινοβούλιο ε, με τη διαδικασία της αναπόφασης σε αυτά τα θέματα. Σε αυτή μου λοιπόν την πρώτη επίσκεψη στην Επιτροπή Ήτρε, νομίζω ότι έχουμε την ευκαιρία να ξεκινήσουμε έναν επικοδομητικό και σε ανοιχτό πνεύμα διάλογο και ελπίζω αυτή η συνεργασία να διατηρηθεί σε όλη τη διάρκεια της θητείας μου. Πιστεύω ότι οι προτάσεις, οι ιδέες σας και οι επικρίσεις σας θα είναι ε, επικοδομητικές και για το πρόγραμμά μας και για τη λειτουργία της αρχής. Βεβαίως, πρώτος και βασικός μου συνομιλητής θα παραμείνει ο κύριος Νίμπλερ, η κυρία Νίμπλερ. Uh, Που είναι βεβαίως εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο και θα εκφράζει τη φωνή του Κοινοβουλίου. Ε, επίσης θέλουμε να έχουμε και ανταλλαγή απόψε μαζί σας για το σύστημα Γαλιλαίου το 2011 θα είναι σημαντικό για το σύστημα αυτό. Να ξεκινήσω από το έγνος. Σε ένα μήνα το έγνος θα κηρυχθεί. Θα είναι μάλλον απολύτως διαθέσιμο για σκοπούς ε, πολιτικής ε, αεροπορίας και τέτοιες χρήσεις. Είναι μια επιτυχία το παράδειγμα του έγνος, έχει δώσει πολύ καλές επιδόσεις και είναι το δεύτερο σύστημα παγκοσμίω μετά το αμερικανικό WASH που έχει βελτιώσει τις επιδόσεις του GPS. Περιμένουμε λοιπόν μέγιστες αλλαγές στη λειτουργία της ε, αεροπλοείας. Θα πρέπει να ξέρετε ότι στις Ηνωμένε Πολιτείε περισσότερες από 500 διαδικασίες έχουν ε, αναπτυχθεί και ελπίζουμε ότι οι προμηθευτές τέτοιων υπηρεσιών στην Ευρώπη πολύ σύντομα θα λάβουν υπόψη αυτές τις νέες γνώσεις για το Γαλιλαίο. Ε, από τις έξι συμβάσεις που ήδη έχουν υπογραφεί υπάρχουν δύο ακόμη που θα περατωθούν μέχρι το καλοκαίρι οπότε καταλήγουμε στο πιο σημαντικό. Το Σεπτέμβριο φέτος η πρώτη δορυφόροι, δύο πρώτοι δορυφόροι, για την προσωμείωση πτήσεων, για την παρουσίαση μάλλον των πτήσεων, θα τεθούν σε τροχιά. Έτσι, από το Σεπτέμβριο θα αναπτύξουμε όλα μας τα δορυφορικά συστήματα. Από αυτή τη στιγμή και μετά θα αποσταλούν στο διάστημα και οι υπόλοιποι δορυφόροι το 2012, 2013 και 2014 και πιστεύουμε ότι οι πρώτοι δορυφόροι σε τροχιά που θα μπορούν να δώσουν τις πρώτες υπηρεσίες θα είναι έτοιμοι το 2014 ή 2015 περίπου. Ε, τώρα η δική μου θεώρηση για το μέλλον, για τον Καλλιλέο. Πιστεύω ότι το δυναμικό που διαθέτουμε ώστε το Galileo μαζί με το GPS να φέρει σε πρωταρχικό ρόλο το σύστημα GNSS και να συμπορευτούν τα δύο συστήματα αυτά ε, είναι κάτι που θα το πετύχουμε με την παροχή υπηρεσιών το 2014 και 2015 και αυτό είναι πρωταρχική σημασία. Πιστεύω ότι το Galileo, το σύστημα, μπορεί να μας επιτρέψει την επίτευξη των στόχων στρατηγικής ανεξαρτησίας και να μας αποφέρει και τα οικονομικά ωφέλη που θέλουμε από το πρόγραμμα αυτό. Σε αυτό το πλαίσιο ε, η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο ιδίως σε δύο τομείς. Από τη μια στην ασφάλεια, ιδιαίτερος για τη λειτουργία των κέντρων ασφαλείας και έπειτα για την πιστοποίηση. Δηλαδή προκειμένου να εγκρίνονται και να ελέγχονται οι προϋποθέσεις ασφαλείας. Ένας άλλος τομέας όπου η αρχή ε, θα συνεισφέρει ιδιαίτερος είναι το κατά πόσον θα χρησιμοποιείται το σύστημα ως εργαλείο. Εδώ στόχος είναι να διαχειριστούμε σωστά τη μεταβατική περίοδο μεταξύ της αποστολής και της χρήσης. Ε, είναι πολύ σημαντικό διότι οι χρήστες του Γκαλιλαίου είναι πολύ και διαφορετικοί. Είναι ένα πρόγραμμα των Γκαλιλαίο που καλύπτει πολλούς διαφορετικούς τομείς. Είναι ένας τομέας σημαντικός αυτός, όπου ελπίζουμε ότι η αρχή μας θα μπορέσει να συνεισφέρει σημαντικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλοί ζήτησαν το λόγο, πρώτος όμως κύριος Κλάντε. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια για τα νέα σας για τα νέα σας καθήκοντα και να περνάτε καλά στην ε, Πράγα. Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να φροντίσουμε ε, να κάτι να κάνουμε για το προσωπικό. άξο ότι υπάρχουν προβλήματα με το προσωπικό της, ε, του οργανισμού αυτού, επειδή η έδρα είναι στην Πράγα κτλ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος Δαρεμέκ. Ε, ε, Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στον εισηγητή. Ξέρετε, εγώ Μένω στη γειτονιά, εκεί, στην Πράγα. Εκεί κοντά στις εγκαταστάσει. Τέλο πάντων, να ρωτήσω κάτι τον κύριο Διευθυντή. Τι θεωρεί ότι είναι το πιο σημαντικό κατά αυτή την πρώτη φάση και για την υπηρεσία και για τον Γαλιλαίο γενικότερα. Και επίσης πώς θα μπορούσε το Κοινοβούλιο να βοηθήσει. Κυρία Τσικάου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον προσκεκλημένο μας ως εισηγήτρια της Επιτροπής Μεταφορών σε ό,τι αφορά τις μεταφορές και το πώς θα καλύπτονται από το πρόγραμμα Galileo και το σύστημα GNSS να επιστήσω την προσοχή σας στο εξής πέραν της ανάπτυξης των υποδομών, που φυσικά θα είναι το βασικότερο στοιχείο, αλλά χρειάζονται και σημαντικές επενδύσεις, μην ξεχνάμε ότι πρέπει να επενδύσουμε και στην έρευνα. Έρευνα για να αναπτυχθούν υπηρεσίες και συγκεκριμένε εφαρμογές. Και αυτό με τέτοιο τρόπο ώστε όταν αρχίσει να λειτουργεί το πρόγραμμα, να λειτουργούν δηλαδή αυτές οι υποδομές, να χρησιμοποιήσουμε ό,τι ήδη έχουμε στη διάθεσή μας, με εφαρμογές και υπηρεσίες που να είναι ήδη έτοιμες, έτοιμες για να συμπεριληφθούν αμέσως στην αγορά. ελπίζω ότι έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα να πείσουμε την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη Έτσι θα έχουμε τους απαραίτητους πόρους για να χρησιμοποιήσουμε το σύστημα GNSS και το πρόγραμμα Galileo ως το δυνατόν περισσότερο. Για την κάλυψη τώρα του GNSS και του EGNOS, στην νοτιοανατολική Ευρώπη και την νότια Ευρώπη, νομίζω ότι αυτά είναι ζητήματα που τα έχετε ήδη σκεφτεί. Αλλά μην ξεχνάτε ότι θέλουμε να έχουμε μια ενιαία αγορά για τις υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τι συχνότητε που θα χρειαστούμε για την σωστή λειτουργία του συστήματο, θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει πρόβληψη. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κυρία Χέρτσοκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πολύ σύντομα να καλωσορίσω και εγώ τον ε, εκτελεστικό διευθυντή της GSA, να σας ευχηθούμε κάθε επιτυχία για το μέλλον και να σας πω ότι σας θεωρούμε στρατηγικό μας σύμμαχο εδώ στο Κοινοβούλιο. Για να μπορέσουμε να πείσουμε την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη ότι αυτές οι νέες τεχνολογίες είναι πραγματικά αναγκαίες. Αναγκαίες για να έχουμε τα αποτελέσματα που Επιθυμούμε στο δυνατόν συντομότερα. Ελπίζουμε να έχετε λιγότερα προβλήματα στη λειτουργία σας. Ε, στην Επιτροπή για τους προπολογισμού εξετάσαμε το ζήτημα όσο πιο ευνοϊκά μπορούσαμε ε, και είδαμε τι γίνεται με τους προπολογισμούς των οργανισμών. Ελπίζουμε με το δικό σας να μην υπάρχουν προβλήματα. Ε, και επίσης θα ήμασταν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι εάν η αρχή σας με τη μέσα που διαθέτει θα μπορούσε να προωθήσει στου Ευρωπαίους πολίτες το προγράμματα αυτά και το σύστημα GNSS ε, κρατώντας τις υποσχέσεις της. Χρειαζόμαστε το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο ε, για να έχουμε τους απαραίτητους πόρους και για τα δορυφορικά προγράμματα και όπως είπε και η κυρία Τσικάου για τις εφαρμογές. Σας εύχομαι λοιπόν κάθε επιτυχία. Μπορείτε να υπολογίζετε, να στηρίζεστε στο Κοινοβούλιο και είμαστε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε μαζί και στο μέλλον ώστε να πετύχουμε ε, τα αποτελέσματα που υποσχεθήκατε στους Ευρωπαίους πολίτες και να μην πάνε χαμένα όσα έχουν ήδη επενδυθεί σε αυτά τα προγράμματα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ντορίντες, θέλετε να απαντήσετε στα σχόλια που έγιναν θα είχαμε ίσως λίγε ε, παραπάνω πληροφορίε έτσι από εσά. Ναι, πρώτα πρώτα, λέει ο κύριο Δεστορίδης, να μην απαντήσω στον κύριο Γκλάντε όσον αφορά την μετακίνηση προς την Πράγα. Δεν το ανέφερα στην ε, εισήγησή μου, όμως νομίζω ότι πρόκειται για ε, μια πάρα πολύ σημαντική πρώτη πρόκληση για την υπηρεσία. Ίσως είναι πολύ νωρίς για να πούμε κατά πόσο είναι η μετακίνηση αυτή. Πρόκειται σε εξάμεινο να έχει υλοποιηθεί. Γιατί θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα τεχνικά θέματα, ε, γιατί θα πρέπει επίσης να δούμε το ότι η ασφάλεια είναι πάρα πολύ βασικό και άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε κατά πόσον ε, η τοποθεσία αυτή ε, θα είναι ό,τι πιο καλό από πλευρά ασφαλείας. Και να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Πάντω, οπωσδήποτε και πάρα πολύ βασικό θα είναι για αυτή την ε, μετακίνηση να κατοχυρώσουμε, να κρατήσουμε την γνώση ε, την εμπειρία που υπάρχει. Αυτός είναι ο πρώτος ε, στόχος μας και οπότε θα πασχίσουμε για να πετύχουμε και κάτι τέτοιο και στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα όσον αφορά την ε, παρατήρηση ε, πάλι που η οποία έγινε όσον αφορά το, το, το, το μέλλον της υπηρεσίας πρέπει να σας πω ότι η συγκρότηση και η λειτουργία του κέντρου ασφαλείας έχουν μπει στην τελική ευθεία. Οπότε και θα ευιστατεύσουμε πάσα προσοχή για να μπορέσουμε να είμαστε σύντονοι με το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει τεθεί, δηλαδή με την καταληκτική κείμενο το 2014. Επίση κύριε Ρέμ, είπατε το ότι θα πρέπει να εξεταστεί το κατά πόσον το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να βοηθήσει την υπηρεσία. Όπως προανέφερα, θεωρώ ότι δυνάμει του νέου εγκριθέντο κανονισμού για πρώτη φορά θα έχουμε εκπρόσωπο του Κοινοβουλίου ή στο Διοικητικό Συμβούλιο. Επομένω, θεωρώ ότι έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε από κοντά τα πραγματικά προβλήματα, τους κινδύνους, τα διαφορετικά θέματα του προγράμματος. Επομένω για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μου πει το Κοινοβούλιο τι κινδύνους επισημαίνεται. Κάτι το οποίο θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο και θα ωφελήσει το πρόγραμμα και την υπηρεσία. Κύριε Τσεκάου, και εσείς τονίσατε το ότι χρειάζεται να επενδύσουμε σε έρευνα ανάπτυξη και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τα θέματα υπηρεσιών, εφαρμογή. Ναι, πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά. Γιατί περίπου 80-90% το, τις του Γαλιλαίου ο, όντως ε, είναι εκεί. Άρα... Εκεί, εκεί, εκεί έγκυται και όχι στην κατασκευή. Επομένως, ε, όλα αυτά πρέπει να τα προσέξουμε. Και έχουμε ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα δράση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο ε, εκεί αφορά τις διαφορετικούς τομείς, κανονισμούς κλπ. Οπότε και θα είναι ε, πρώτος μου στόχος για να συνεργαστούμε με την Κομισιόν και να υπάρξει ένα τέτοιο σχέδιο δράσης. Εγώ θα πρέπει να παραδεχτώ ότι υπάρχει ένα σημαντικό θεματάκι. Ακριβώς η έλλειψη χρηματοδότησης όσον αφορά το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο τελευταία, όσον αφορά την δημοσιονομική προοπτική. Είναι πάρα πολύ περιορισμένα τα πράγματα, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο ε, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση κατά την οποία Φαρμαγέ υπηρεσίε δεν χρηματοδοτούνται ακριβώς σε μια συγκυρία κατά την οποία χρειάζεται περισσότερο. Επομένως τώρα εδώ θα πρέπει και να μοχλεύσουμε. Να ανακινητοποιήσουμε ό,τι, ό,τι είναι δυνατόν να υπάρξει. Αφρυπίν. Ε, συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τραπεζα Επενδύσεων, να βρεθούν τα κατάλληλα μέσα, ούτω ώστε να μπορέσουμε και να κάνουμε αυτό που πρέπει. Κάτι τελευταίο με προποθετικό αυτό το οποίο αναφέρατε για το σύστημα έγνος ότι όντως έχετε δίκιο στην Ανατολική Ευρώπη υπάρχουν κάποια θέματα για την κάλυψη αλλά Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι γνωστό και θα αντιμετωπιστεί και είναι πάρα πολύ βασικό για την ε, Κομισιόν. Και θα μπορέσουμε και θα καλύψουμε και τις υπόλοιπες χώρες τελικά. Κάτι άλλο τώρα. Σαν φορά τις συχνότητες. ο Γαλιλαίος εδώ. Είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει διαλειτουργικότητα πλήρης με το GPS, κάτι το οποίο αποτελεί ένα τρομερό πλεονέκτημα όσον αφορά τις συχνότητες, κωδικούς, κώδικες πρόσβασης, ε, formatting των δεδομένων, αυτό σημαίνει διαλειτουργικότητα και επίσης ε, ακόμα και αν δεν έχουμε όλο, όλο το, το, το, σχηματισμό σε ανάπτυξη. παρόλα αυτά ε, πρόκειται για αξιοποίηση των υπηρεσιών γιατί σήμερα αυτή η διαλειτουργικότητα ε, δεν είναι αυτονοητή ούτε για το ρώσικο ούτε για το σύστημα το κινέζικο. Επομένως πρόκειται για ένα τούτο το οποίο θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Επίσης, τώρα πολύ συγκεκριμένα, όσον αφορά τις ε, δημόσιες υπηρεσίες, εκεί όπου ας πούμε οι, οι συχνότητες ε, είναι κινέζικες κλπ. Και το, το, το οποίο αντιμετωπίζει η Κομισιόν. Τώρα. Τελευταίο. Τελευταία παρέμβαση αφορούσε το, το μέλλον της υπηρεσίας. Και ότι δεν είναι επιθυμητό να έχουμε και πάλι κάποια προβλήματα τα οποία είχαμε στο παρελθόν στην υπηρεσία. Επομένως γι' αυτό και πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία δύο χρόνια τα έχω περάσει σε, στην Κομισιόν, εκεί δουλεύω. Επομένως ελπίζω ότι εδώ πέρα έχω κάτι να εισφέρω και θεωρώ ότι υπάρχει σχέση σημαντική με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο είναι ένα πλεονέκτημα. Βεβαίως, λαμβάνοντας υπόψη και την ε, καινούργια υπηρεσία, αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, κατακλείδη, να σας πω ότι πρόσφατα έχουμε την έκθεση Ταγιάννη. Θα συζητήσουμε στο την προηγούμενη εβδομάδα για αυτή τη μεσοπρόθεσμη ε, αναθεώρηση, οπότε ανοιχτή πια η συζήτηση σε κοινοβούλιο και συμβούλιο σε όλο το μέλλον του Γαλιλαίου και είναι πάρα πολύ σημαντικό ζητήματα αυτά και μιλούμε για την ε, μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και την διακυβέρνηση. Μπορώ να σας πω ότι θα κάνω ότι περνάει από το χέρι μου γιατί θεωρώ ότι η συνεργασία και η εκμετάλλευση του Γαλιλαίου θα πρέπει να γίνει από αυτή την καινούργια υπηρεσία, την οποία και εγώ θα υποπτεύω και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όλος που έχω να διαδραματίσω. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κύριε Ντορίδης εκ μέρους της Επιτροπής για την ε, παρουσία σας εδώ. Θα ήθελα να σας πω επίσης ότι ε, πράγματι πιστεύω ότι θα συνεργαστούμε καλά, ιδιαίτερα οι συνάδελφοι που είναι αρμόδιοι και υπεύθυνοι για τα θέματά σας. Ζητώ συγγνώμη για σήμερα, έπρεπε λίγο να βιαστούμε, αλλά είχαμε πρόβλημα χρόνου. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που ήρθατε, σας εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες σας και εύχομαι και καλή συνεργασία ε, με την Επιτροπή μας. geht direkt in die Debatte weiter. Darf bei uns Herr Minister Schäfer. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον ε, Υπουργό Τζεφαλκβάη. ελπίζω να πρόφερα σωστά το όνομά του είναι υφυπουργό στρατηγικών υποθέσεων αρμόδιο για τη βιομηχανία και την έρευνα και άρα είναι και πρόεδρος του Συμβουλίου των Υπουργών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Α μην χάσουμε το χρόνο μας με εισαγωγέ δικέ μου θα δώσω κατευθείαν το λόγο στον ε, Υπουργό του ώστε να έχουμε χρόνο και όλες μετά να συζητήσουμε να κάνουμε εκτενή συζήτηση πριν δούμε τις λεπτομέρειες για να δούμε ακριβώς τι διακυβεύεται εδώ που συζητάμε για βιομηχανία και έρευνα στην Ευρώπη. Έχουμε αντιλήσει κάποια συμπεράσματα, έχουν πάρει το μάθημά μας και τώρα ήρθε η ώρα κάτι να κάνουμε με αυτά τα μαθήματα γιατί έχουμε αυτή την ε, συνεργασία όσον αφορά και δημοσιονομική πολιτική και έχουμε τώρα τη χρηματοπιστωτική πολιτική. Έχουμε φτάσει σε κάποιες ανισορροπίες όμως θεωρώ ότι υπάρχουν κάποια άλλα θέματα τα οποία είναι σημαντικά αλλά είναι λιγότερο φανερά. Να σας πω τι σκέφτομαι. Οπότε απλώς και επισύρω την προσοχή σας στα εξή τρία ζητήματα. Μα απασχολεί η διαχείριση τη κρίση και η σταθερότητα, αλλά να μην ξεχνούμε ότι θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειε για την ανταγωνιστικότητά μα. Και εμεί πιστεύουμε ότι αν η ανταγωνιστικότητα δεν σιγουρευτεί, αν δεν φτάσουμε σε μεγαλύτερη ανάπτυξη, δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα δημοσιονομικά. Δεύτερον, ε, υπάρχουν όλο ένα και περισσότερα σημάδια για το ότι ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό το να αντιμετωπίσουμε την κρίση με την καινοτομία. Και έτσι θα πάνε καλύτερα και οι επιχειρήσεις στην καθημερινή του λειτουργία, αλλά αυτό αφορά και πολιτικέ φιλικές στο περιβάλλον. Επίσης δεν θα πρέπει να ξεχνούμε το ότι θα πρέπει να έχουμε αηφόρο ανάπτυξη και ότι θα πρέπει να έχουμε δημιουργία εργασία. Γιατί ανάπτυξη χωρί θέσει εργασία καινούργιε δεν ωφελεί να δώσουμε κάποια συμπεράσματα από την κρίση. Τα οικονομικά προβλήματα έχουν τη ρίζα τους σε αίτια πολιτικά, στους ανθρώπινα κουσούρια και όχι σε οικονομικά ζητήματα. Άρα χρειάζονται αντίστοιχες ε, απαντήσεις από τα κρατημέλη αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση επομένω. Θα πρέπει να δούμε το τι χρειάζεται, να δούμε πώς θα πρέπει να δούμε το σύνολο του τοπίου. Να δούμε και τις λεπτομέρειες επομένω και το σύνολο και το δέντρο και το δάσος, οπότε και έτσι μπορούμε να δούμε το θέμα της πολιτικής με το 2020, κάτι το οποίο δεν είναι απλώς μια διάδοχη κατάσταση της Συνήθλης Λισαβόνας. Είναι μια πολιτική η οποία θα μας οδηγήσει να δούμε στο τι διακυβέρνηση θα ασκήσουμε και πώς θα έχουμε κάποιο είδου ε, μεταρρύθμιση της πολιτικής μας σε ευρωπαϊκό και κρατικό επίπεδο. Επίσης θα πρέπει να δούμε ποιος θα είναι ο χάρτης πορείας για να έχουμε μια καινούργια διάσταση, μια οικονομική εποπτεία και συντονισμό. Το ΕΚΟΦΗΝ βέβαια έχει τον βασικό πρωτοδομιστικό ρόλο, όμως ε, και αλλού στο Συμβούλιο πολλά μπορεί να γίνουν. Γι' αυτό σας λέω ότι το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας επίσης πρόκειται να τα συζητήσει. Και εδώ πέρα το θέμα είναι να έχουμε κάποια συνοχή, πρωτοβουλίες, καινοτομία και ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική. Επίσης βλέπουμε εδώ ένα σωρό θέματα. Πολλά από αυτά εκκρεμούν πολύ καιρό και κάποια όμως αφορούν πρόσφατες εξελίξεις οι πολίτες και οι επιχειρήσεις περιμένουν από μας να βρούμε ένα διέξοδο στα διέξοδα. Να δούμε πώς θα δοθούν καινοτόμες λύσεις στις πρόσφατες προκλήσεις. Σε τρεις άξονες ε, θα κινηθεί το Συμβουλίο Θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε τόσο ώστε να πάει σε ανάκαμψη η Ευρώπη. Θα πρέπει επομένω οι επιχειρήσει να είναι λιγότερο θα πρέπει να έχουμε λιγότερου φραγμού, θα πρέπει να είναι δυνατόν οι εταιρείε να μπορούν να λειτουργήσουν με λιγότερα έξοδα σε πανευρωπαϊκή κλίμακα. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από την ε, κρίση, να έχουμε ανάπτυξη, να δημιουργήσουμε θέσει και αυτό που χρειάζεται τώρα δεν χρειάζεται πολυνομία μεγαλύτερη. Το αντίθετο, θα πρέπει να άρουμε του περιορισμού. Οπότε υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία ε, θα πρέπει να τα δούμε, έντυπα διοικητικές δαπάνες, όλα, όλα αυτά τα έξοδα. Γιατί αυτά όλα κοστίζουν σε πόρους, σε αποτελεσματικότητα, επομένως θα πρέπει ε, οι λαμβάνοντες αποφάσεις να αναρωτηθούν. Και εδώ πέρα έχουμε ένα σωρό ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Πολύ σημαντικό θέμα είναι η πράξη για τις ΜΜΕ, δημιουργία θέσεων εργασίας, ε, παραγωγή, όμως οι ΜΜΕ πέραν αυτών παλεύουν να βρουν χρηματοδότηση, δεν έχουν εσωτερήκευση των εξόδων και ο λόγος είναι η ίδια τους η φύση. το πρόβλημά τους. Δεν είναι το μέγεθός τους. Αλλά το ότι δεν μπορούν να επηρεάσουν τα πολιτικά δρόμενα, το πολιτικό περιβάλλον και το αριθμιστικό περιβάλλον. Γι' αυτό. Είναι μοναχικοί καβαλάριδες και αυτό θα πρέπει να έρθει. Επομένως, να τις βοηθήσουμε με λιγότερη γραφειοκρατία. Να μπορούν να έχουν προσβασιμότητα σε ξένε αγορέ και στην καινοτομία επίσης να έχουν πρόσβαση. Να τις βοηθήσουμε να μεγαλώσουν, να δυναμώσουν. Ο Σούμαχερ είπε το περίφημο το μικρό είναι όμορφο αλλά εγώ σας τονίζω ότι θα πρέπει με τις πολιτικές μας να βοηθήσουμε τις ΜΜΕ να μεγαλώσουν να του επιτρέψουμε, να του αφήσουμε μεγάλου γιατί μπορεί το μικρό να είναι όμορφο, αλλά το να δυναμώνει ο μικρό είναι ακόμα πιο ελκυστικό. Να μπορούν να πάνε σε αγορέ, να δώσουμε χρηματοδότηση, να πλουστεύσουμε το νομικό περιβάλλον. Εμείς στην Προεδρία μας θα χρησιμοποιήσουμε την ε, μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση και επίσης περιμένουμε το ιερινό έγγραφο της Κομισιόν. Το Μάιο θα βγουν κάποια συμπεράσματα και εκτός από τη, τα, επίσημα συνέδρια εμείς θα έχουμε σε επαφή με τους συναρμοδίους υπουργού άτυπα και έτσι θα είμαστε σε επαφή για να μειώσουμε τα διοικητικά, να μειώσουμε την κρατική, τις κρατικές ενέργειες, ε, να έχουν μεγαλύτερη παραγωγική δυνατότητα οι ΜΜΕ, αυτό να μπει στην ε, πράξη για τη ΜΜΕ. Σωτερή των τον επίσης των ΜΜΕ. Εκτός, επομένως, από τις άλλες εκδηλώσεις θα έχουμε 24 και 25 Μαΐου μια, ένα συμπόσιο για τις ΜΜΕ. Θα βραβεύσουμε την επιχειρηματικότητα, τις καλύτερες πρακτικές. Βεβαίω και το κόστος της συναλλαγής είναι πολύ σημαντικό. Όμως, όσο υπάρχει κατάτιμη στην αγορά και όσο υπάρχει προβλήματα στην κινητικότητα, ακόμα δεν μπορούμε να αυτό το οποίο θέλουμε πάνω αυτό το οποίο θέλουμε. Είναι να βρούμε κάποιες πολιτικές, ούτω ώστε να καταπονημήσουμε αυτές τις στρεβλώσεις και να μπορέσουμε να έχουμε κινητικότητα παντού. Το είπε ο Άνταμ Σμιθ ότι η παραγωγικότητα και οι θέσει απασχόληση προέρχονται από την κατανομή εργασία. Αλλά βέβαια αυτό εξαρτάται πάλι και από την ε, αγορά. Άρα αυτό είναι εφικτό όταν μπορούμε να φρενάρουμε την ε, κατάτμιση της αγοράς που φέρνει ε, υπερβολική δύναμη της αγοράς, αποτρέπει τις επιχειρήσεις να έχουν οικονομίες κλίμακος, εμποδίζει τις επενδύσεις θέση απασχόλησης και επομένως η κατάτμιση της αγοράς σημαίνει ότι μειώνονται δυνατότητες για την οικονομική ανάπτυξη και θα πρέπει μένως αυτοί που χαράσουν την οικονομική πολιτική πάντοτε να αναρωτιόνται αν όντω καταπολεμούν την κατάτμιση και αν βοηθούν τις επιχειρήσεις. Να σας πω τώρα τι θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ερευνητική περιοχή στην Ευρώπη απεδείχθη πολύ καλή ιδέα, όμως τα εθνικά και το ευρωπαϊκό σύστημα, η ευρωπαϊκή διάσταση, είναι πράγματα τελείως χωριστά τώρα και γι' αυτό και έχουμε έξτρα κόστος και επικαλύψεις. Επομένως, για να αντιμετωπίσουμε την κατάτιμηση, θα προσπαθήσουμε να κατατείνουν στο να βοηθήσουμε το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και γι' αυτό ακριβώς έχουν χρησιμοποιήσει αυτών των ε, ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων με τους οποίους είμαστε σε επαφή και εγώ επομένως επειδή με αυτό έχω ασχοληθεί έχω ευαισθησία για το θέμα οπότε και πιστεύω θα πρέπει η Ευρώπη να φροντίσει σε όλες τις πτυχές την ε, έρευνα επιστήμη, κοινωνία, ανταγωνιστικότητα, ούτω ώστε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Ρίξτε μια ματιά στην ενδιάμεση έκθεση και θα δείτε ότι περιέχονται εκεί 10 συστάσεις. Οπότε εδώ έχουμε το ποιοτικό άλμα. Και κατά τη γνώμη μας η καινοτομία οδηγεί σε καλύτερη διοίκηση. Τώρα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά αυτές τις στάσεις, γιατί νομίζουμε ότι έτσι θα ανοίξει ο δρόμος για συμμετοχή των κρατών μελών, που τώρα υποεκπροσωπούνται. Να καλύψουμε και τις χώρες κεντρικής και κεντρικής Ευρώπης, για μια ματιά στα στοιχεία. τον πληθυσμό, κοιτάξτε, και τις άλλες μεταβλητές. Οπότε θα κάνουμε και αυτή τη διάσκεψη όσον αφορά την 24η-25η Φεβρουαρίου. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τις συστάσεις. Στο πλαίσιο του εβδόμου, πρόγραμμα προγράμματος πλαίσιου. Θα γίνει η ανταλλαγή απόψεων τον Μάρτιο και καταλήξω κάποια συμπεράσματα πάντως. Ρίξτε μια σε αυτές τις 10 συστάσεις και θα δείτε ότι εδώ πέρα υπάρχουν προτάσεις για το μέλλον. Να σας αναφέρω τρεις. Το επίπεδο της χρηματοδότησης θα πρέπει να είναι το ίδιο. Ξέρω ότι αυτό θα προκαλέσει ζωντανές συζητήσεις στο μέλλον. Αλλά αυτό έχουν πει οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες τώρα. Θα πρέπει να υπάρχει διαφορετική προσέγγιση. Και αυτό και θα κάνουμε στο Ιαρινό Συμβούλιο τον Απρίλιο. Να δούμε δηλαδή πώς θα είναι η διαφορετική προσέγγιση για το πρόγραμμα πλαίσιο να είναι λιγότερες οι δαπάνες για τη λειτουργία τη επιχείρηση. Να είναι στην παγκοσμιωμένη αγορά πιο πετυχημένες επιχείρησεις μας. Γι' αυτό και χρειάζονται κάποιες κοινωνικέ πολιτικές για περισσότερη ανταγωνιστικότητα τη βιομηχανία και των επιχειρήσεων παντού στον κόσμο. Παρά το ότι είμαστε καλοί στην ανώτατη εκπαίδευση, εμείς στην καινοτομία δεν τα πάμε τόσο καλά, δηλαδή πόση έρευνα θα αξιοποιείται. Αν το δούμε αυτό στα πλαίσια του 2020 θα πρέπει να συντονίσουμε τις προσπαθίε μας. Και ξέρετε τι πει η Αγγέλα Μέρκελ. Η ευημερία μας μπορεί να συνεχιστεί μόνο εάν συνεχίσουν να είμαστε καινοτόμοι και πρωτοπόροι. Θα πρέπει να δούμε και οι πόροι θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις. Γι' αυτό και η σχετική πρωτοβουλία είναι πάρα πολύ σημαντική. Να γίνει προτεραιότητα το Συμβούλιο. Κατέληξε σε συμπεράσματα και θα πάρει τη τώρα η Ουγγρική Προεδρία και είναι πάρα πολύ σημαντική η προτεραιότητα τώρα υπάρχει εταιρική σχέση εδώ και αυτή η συνεργασία να έχει πιλωτικό χαρακτήρα. Οπότε και το Ίδρυμα για Καινοτομία και Τεχνολογία επίσης έχει να παίξει σημαντικό ρόλο. Είναι στατική σημασία η ατζέντα που αφορά τα θέματα της καινοτομία επίσης. Οι κοινέ πρωτοβουλίε πάλι είναι σημαντικές για την έρευνα. Οπότε και αυτά θα είναι απόσπασμα της στρατηγικής του 2020. Σχοληθούμε και με τις πρώτες ύλε. γιατί θεωρούμε ότι έτσι θα έχει περισσότερη αυταργία ασφάλεια προσφορά η Ευρώπη. Έχουμε το πρόγραμμα δράσης που θα υλοποιήσει αυτές τις ε, προτεραιότητες ανάλογα με το τι θα αποφασίσει το Σύμβουλο Ανταγωνιστικότητας στην Άνοιξη. Κυρίες και κύριοι, η Ευρώπη σήμερα έχει αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις, θα απαιτήσουν μεγάλες προσπάθειες από όλους. Η φιλοδοξία μας είναι βέβαια να γίνει ισχυρότερη η Ευρώπη. Αυτό είναι το σύνθημα της ε, Ουγγρικής Προεδρίας. Η Ένωση ανήκει σε όλα τα μέλη και θα πρέπει να την κατοπτρίζει τις παραδόσεις του κάθε μέλους και αυτό το είπε η Μάργαρη Θάτσα, δεν το έχω πει εγώ. Γι' αυτό και νομίζω ότι θα πρέπει να διευρύνουμε τον οριζοντά μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανήκει σε όλους τους πολίτες Άρα θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τι προσδοκίε των πολιτών. Οπότε νομίζω ότι το Συμβουλίο Κοντές και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συνεργαστούν στενά και τότε έχουμε πάρα πολλέ φάνατες να ξεπεράσουμε τι δυσκολίε. Να είναι λιγότερο δαπανηρή η δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Να σταματήσουμε την κατάρτιση αγορά και όσον αφορά την έρευνα και επίση να γίνει πιο μεγάλη, πιο καλή ένταγωση των επιχειρήσεων. Αν κάνουμε αυτό το οποίο μα αναλογεί, θα πετύχουμε την ανάκαμψη. Ευχαριστούμε του προκατόχου μα, το Βέλγιο, την Ισπανία και του άλλου. Και όσον αφορά την ε, βιομηχανία και έρευνα, μα βοήθησαν πάρα πολύ και εμεί είμαστε δεσμευμένοι, υποσχόμεθα να συνεχίσουμε στο ίδιο πνεύμα σε στενή συνεργασία μαζί σας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ούτως ώστε με τις επόμενες πρωτεύουσες Πολωνία και Δανία να συνεργαστούμε. Σας ευχαριστώ πολύ την προσοχή σας και με μεγάλη ευχαρίστηση να απαντήσω στις τυχόν Ευχαριστώ πολύ. Ήδη έχουν ζητήσει πολύ το λόγο. Ε, ένα λεπτό δίνω για τις ερωτήσεις. Ο κύριος Κιούκ είναι ο πρώτος. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ για την εισαγωγή κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα να πω πρώτα πρώτα ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που η Ουγγρική Προεδρία ε, βλέπει όχι μόνο τα δέντρα αλλά και το δάσος και χαίρομαι ιδιαίτερα που θα ασχοληθείτε και με θέματα έρευνας ε, ε, ακόμη και σε χρόνους ε, οικονομικής κρίσης. έρευνα και καινοτομία είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη τα οποία ε, δεν προχωρούν με τον ίδιο τρόπο και δεν ναι, εκπροσωπούνται με τον ίδιο τρόπο στα μεγάλα προγράμματα ως τα μεγάλα κράτη-μέλη ας πούμε. Παρακαλώ. Ναι, ναι, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που αναφερθήκατε ε, τόσο πολύ στην ε, καινοτομία. Ε, εγώ όμω θέλω να ρωτήσω... Uh, θα ήθελα να μου πείτε πώς συνδέεται και το καινοτομία με αυτό που ορίζεται ως analog hard economy. Από εκεί και πέρα ο Μίλτον Φρίντμαν είπε ότι there is no such thing as a free lunch. Οπότε ε, ε ποιος κερδίζει από αυτή την υπόθεση. Και από εκεί και πέρα ε, όλοι μιλούμε για εμπιστοσύνη, δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης αλλά ο Έρχαρτ είχε πει παλιά ότι η εμπιστοσύνη είναι καλό πράγμα αλλά ο έλεγχος απαραίτητος λοιπόν ε, τι λογοαριάζεται να κάνετε σχετικά και ούτως ή άλλως αναφερθήκατε βέβαια με αρκετό λυρισμό και ρομαντισμό στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Από εκεί και πέρα ε, είπατε ότι θα δώσετε στοιχεία ήδη από το Μάιο. Πώς θα, τα κατα... έχετε κα... αποτελέσματα ήδη το Μάιο. Πώς θα τα καταφέρετε κυρία Καβάλιο. Ευχαριστώ. Ήθελα να πω ότι ελπίζουμε πολλά από τη δική σας Προεδρία και χαιρόμαστε που προβλέψατε τη διαδικασία την απλουστευμένη και για την κοινοτομία. Ε, εδώ το Κοινοβούλιο πρόσφατα ενέκρινε μια πρόταση για την διαδικασία απλούστευσης στα προγράμματα έρευνα και καινοτομία. Είναι σημαντικό το, είναι σημαντική η δέσμη μέτρων ε, της Επιτροπής. Τώρα Βλέπουμε ότι έχουμε περάσει τη φάση υλοποίηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά έχουν παραμείνει κάποια προβλήματα και τα έχει εντοπίσει και το Συμβούλιο. Όχι το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητα, η Υπουργή Οικονομικών. Για το ανεκτό επίπεδο σφάλματος, ε, Υπουργέ, πώς θα μπορούσαμε να προωθήσουμε περαιτέρω τη διαδικασία απλούστευση. Ευχαριστούμε κυρία Χέρτσοκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είστε ο πρώτος, κύριε Υπουργέ, που χειροκροτήθηκε εδώ στην Επιτροπή μας. Θα ήθελα κι εγώ να σας συγχαρώ για αυτά που είπατε. Αλλά κατά κύριο λόγο να ρωτήσω κάτι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ξέρω ότι αυτές οι επιχειρήσεις είναι υψηλή, χαίρουν υψηλής προτεραιότητας με εξωθωμάτων της Ουγγρικής Προεδρίας. Καταλαβαίνουμε και εμείς τις δυσκολίες και πιστεύουμε ότι ένα από τα σοβαρά ε, θέματα είναι όχι η πρόσβαση σε, ε, στα κεφάλαια, αλλά η χρέωση, τα χρέη που κάνουν επιχειρήσεις αυτές. Επίσης, εσείς μιλάτε για καινοτομία, για ψηφιακές τεχνολογίες που θα πρέπει να απορροφηθούν και να χρησιμοποιηθούν και από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όλα αυτά τα πράγματα όμως κοστίζουν, δεν ε, έχουν τον εξοπλισμό οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα πρέπει να δανειστούν για να τα για να εξοπλιστούν αντίστοιχα. Χαίρομαι που προς το τέλος Μαΐου θα οργανωθεί και πάλι μια ε, συνδιάσκεψη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα ήθελα όμως να μου πείτε γιατί δεν γίνονται άλλες συνεδριάσεις που τις αναλαμβάνει τώρα η Πολωνική Προεδρία ενώ πρώτα γινόντουσαν κάθε εξάμεινο. Κύριε Υπουργέ, έχετε τώρα εσείς το λόγο, μπορείτε να απαντήσετε. és a, a fát, ami ennyi dossziénél nem egy Ναι, κάποιος είπε ότι βλέπουμε ότι το δάσος και όχι μόνο τα δέντρα. Όντως ε, θα πρέπει να βλέπουμε και τα επιμέρους αλλά και το γενικό πλαίσιο και τη γενική ατμόσφαιρα. Πραγματικά νομίζω ότι δεν είναι δυνατόν να αγνοούμε το γενικότερο περιβάλλον. Ανέκαθεν αυτό έκανα και αυτό θα συνεχίσω να κάνω και ως πρόεδρος του Συμβουλίου εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, για την ενδιάμεση έκθεση σχετικά με το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο είναι γεγονός ότι τα ερευνητικά ιδρύματα ιδιαίτερα στην ε, ορισμένα ερευνητικά ιδρύματα έχουν μικρότερες δυνατότητες να χρηματοδοτηθούν από την Ένωση από τι άλλα ήρθα σε συνεργασία με ένα συνάδελφο από το LSE ε, καθίσαμε και, και μελετήσαμε λιγάκι το θέμα είδαμε ότι με, μελετήσαμε τη μετά, την εποχή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και είδαμε ότι έγιναν πολλές, σε πολλές χώρες πολλά και σημαντικά λάθη. Άλλες, αλλού όμως και σε άλλες χρονικές στιγμές έγιναν πολλά θετικά πράγματα. Αυτή τη στιγμή το κύριο πρόβλημα είναι ότι ίσως ελείπει η υποδομή. Δεν υπάρχει υποδομή για να στηρίξει τους ερευνητές. Και αυτό πρέπει να ε, συζητήσουμε νομίζω. Πώς μπορούμε να αναπτύξουμε τις υποδομές ούτως ώστε η εργασία των ερευνητών να διευκολυνθεί. Μην ξεχνάτε, στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο η λέξη κλειδί είναι η αριστεία και θέλουμε να συνεισφέρουμε κι εμείς να δημιουργηθεί η αριστεία και τα δίκτυα αριστείας. Φαίνεται πως στις ε, ανατολικές ευρωπαϊκές χώρες μπορεί να υπάρχουν τα κονδύλια τα οποία θα δοθούν από κάπου αλλά οι υποδομές δεν υφίστανται δείτε πόσο είναι το ποσοστό των επιτυχών προτάσεων που υποβάλλονται 15 με 20% και βεβαίως δεν μπορούν να είναι όλοι άριστοι αυτό είναι γεγονός αλλά το ποσοστό των αυτών που κερδίζουν προγράμματα είναι το ίδιο στην Ανατολική και στη Δυτική Ευρώπη ωστόσο άμα δεν υπάρχει η, σο η, η υποδομή στην Ανατολική Ευρώπη τότε τα πράγματα δεν πάνε καλά τώρα συνεχίζω στα γερμανικά το όρος καινοτομία είναι ένα ιδιαίτερα αγαπητός όρος και ένα ιδιαίτερα αγαπητό θέμα το οποίο θα προωθήσουμε. Δεν Θέλουμε όμως, που δεν είναι λόγο όμως, η καινοτομία θα πρέπει να σημαίνει γραφειοκρατία. Δεν θέλουμε να περνάμε την ώρα μας να συμπληρώνουμε έντυπα και οι επιστήμονες πολλές φορές όταν βλέπουν αυτές τις ε, τεράστιες γραφειοκρατικές διαδικασίες στη φάση της προετοιμασίας κόνουν χέρια ψηλά και δεν συμμετέχουν. Λοιπόν, ε, αυτή Επίσης λάβετε υπόψη ότι στην ε, κεντρική και ανατολική Ευρώπη δεν υπάρχει και η διοικητική στήριξη, η γραμματιακή στήριξη που υπάρχει στο, στην ε, Δυτική Ευρώπη και είπατε είπατε ότι there is no such thing as a free lunch. Ε, δεν είναι του Μίλτον Φρίντμαν αυτό. Η... Και η φράση δεν ήταν πλήρη που είπατε. Είπατε ότι ε, πρέπει να συμπληρώσετε με το άλλο κομμάτι που λέει ότι ακόμη και αν υπάρχει, όταν υπάρχει free lunch, η τιμή του ή το τίμημα γι' αυτόν διπλάσιο από ό,τι διαφορετικά. Λοιπόν, τέλο πάντων, δεν θέλουμε να πληρώσουμε με άλλα λόγια ε, το τίμημα της γραφειοκρατίας για να προωθήσουμε την καινοτομία. Ναι, αλλά η διαφορά μεταξύ έρευνας και καινοτομίας και χρηματοδότησης έρευνας και, τε, ε, και καινοτομίας, αυτές οι διαφορές παραμένουν, ε, βεβαίως παραμένουν, λέει ο κύριος Κεφαλβάη παραμένουν διότι θέλουμε να υπάρχουν ε, για την έρευνα χρήματα στο Ταμείο για να μπορέσει να προωθηθεί η γνώση. Η καινοτομία είναι χρήματα που διατίθεται για να δημιουργηθούν πηγές χρήματος και πάλι, ε, επιχειρηματικότητα κτλ. Simplification, ich uh... Απλούστευση. Ε, έχουμε μια ομάδα εργασία όπου οι υπουργοί ασχολούνται με τα μέτρα εργασία. Θα έχουμε λοιπόν μια πολύ συγκεκριμένη λύση για το πώ μπορούν να προχωρήσουν όλα αυτά. Ακολουθούμε την προσέγγιση των τριών προεδριών και ελπίζω ότι το Συμβούλιο θα τα αντιμετωπίσει με συγκεκριμένα μέτρα, με προτάσεις για συγκεκριμένα μέτρα για την απλούστευση της όλης διαδικασίας. Τελευταία ερώτηση νομίζω ήταν Σχετιζόταν με, τη, το, τα χρέη των επιχειρήσεων μεταξύ τους, αν θέλετε, και όχι σε σχέση με το δημόσιο. Νομίζω ότι το θέμα αυτό πράγματι πρέπει να μας απασχολήσει και είναι στα διάφορα κράτη-μέλη πρέπει να γίνουν προσπάθειες για να εφαρμοστούν κάποιες νομιού διατάξεις που υπάρχουν ήδη σχετικά με αυτό. Τώρα, όσον αφορά την Ουγγρική Προεδρία, όντω θα δώσουμε υψηλή προτεραιότητα στα θέματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θέλουμε να μειώσουμε το γραφειοκρατικό φόρτο που υπάρχει για τις επιχειρήσεις αυτές. Δυστυχώς δεν είναι εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Τώρα, για την εβδομάδα που γινόταν στο παρελθόν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και που τις αναλαμβάνει τώρα να την οργανώσει, η Πολωνική Προεδρία λυπάμαι και εγώ, αλλά δεν είχαμε χρόνο να την οργανώσουμε στην Εκλογική Προεδρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που ήρθατε, μας δώσετε πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Ε, σας ευχαριστώ που καταφέρατε, βοηθήσατε κι εσείς, ούτω ώστε να καταφέρουμε να τελειώσουμε σύντομα. Και... με, μας, με εντυπωσίασε και εμένα και φαντάζομαι και άλλους συναδέλφους στο γεγονός ότι μπορείτε άνετα να χρησιμοποιείτε τόσες ξένες γλώσσες. Λοιπόν, ελπίζουμε να τα ξαναπούμε. Σα ευχαριστούμε που ήρθατε. Λίγη συνεδρίαση. Σα παρακαλώ να φύγετε ε, ήρεμα και γρήγορα όμως από την αίθουσα γιατί έχουμε συνάντηση των συντονιστών.